Bueno, vayan tomando asiento, por favor. Quiet, please. Ah Vienen, vamos. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τη συναντήρια της Επιτροπής. Έρχεται μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας. Bien. Καλώς. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Μαυρτανίας για τις αλληλευτικές δυνατότητες ε, και ε, την ε, συμφωνία που έχει καθοριστεί μεταξύ των δύο μερών. Έχετε τον κατάλογο των ψηφοφοριών, είναι μία πολύ απλή ένερη διαδικασία όπως γνωρίζετε, δύο τροπολογίες υπευλήθησαν και κατόπιν έχουμε το κείμενο του συντάκτη της σύστασης. Θα ψηφίσουμε λοιπόν καταρχάς τις τροπολογίες. Ε, έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες της κυρίας Λεβίν και του κυρίου Αρσένη. για να εγκριθεί η συμφωνία. Καταρχάς λοιπόν ψηφίζουμε τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τερμίνα. Πέρασε της ψηφοφορίας. 9 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία περιθμών 3. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την νομοθετική πρόταση όπως την είχε υποβάλει ο συντάκτης της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε η ψηφοφορίας. Υπέρ 16, 6 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. θα έλεγα συγχαρητήρια στον υποφαινόμενο, αλλά δεν θα το πω. Έτσι θα πω σκέτο στον ε, συντάκτη της νομοδότησης. Συγχαρητήρια λοιπόν. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Ησυχία παρακαλώ γιατί ψηφίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Προϋπολογισμός 2014. Ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προϋπολογισμός 2014. Εντολή για τον τριμερή διάλογο συντάκτης της νομοδότησης ο κύριος Ριβελίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Οκτώ ψήφοι υπέρ, ε, 10 κατά, απορρίπτεται η πρόταση. Τροπολογία υπαριθμών 3, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 2, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Άρχεται ψηφοφορία. Τροπολογία 10 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. σε δύο τμήματα, συγγνώμη. Το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα, πέραση ψηφοφορία, ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Απροβάδο. Φελικιδάδες. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ριβελίνη. Bueno, finalizadas las votaciones. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Τροποποίηση του κανονισμού 812-2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεπίπτοντα αλλιεύματα κοιτοϊτών κατά την αλληλεία για την τροποποίηση του κανονισμού 88 98. Πρέπει να ψηφίσουμε Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο για να ξεκινήσει επισήμως διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εγκρίνει την ε, επίσημη εντολή. Μην φεύγετε γιατί πρέπει να ε, ψηφίσουμε και μάλιστα ε, με απόλυτη πλειοψηφία. Μαρία, μην φεύγετε. Ένα λεπτάκι να ψηφίσουμε. Είναι απλώς η εντολή για την θέση την οποία θα τηρήσουμε κατά την πρώτη ανάγνωση για να μπορέσουμε να το υποβάλουμε και στην Ολομέλεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Αποχές. Καμία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την εντολή. Uh, without Ψήφισαν όλοι. Οκ. Bien, votos. Termina la votación. Ωραία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν μία ψήφος κατά μόνο. Απόλυτη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 14, ενημέρωση σχετικά με τους τρισμερείς διαλόγους. Έχουμε δύο εκθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να ε, κάνουμε, δύο αναφορές. Ε, το ένα για το βασικό κανονισμό, ε, εκθέση Ρόντουστ και έκθεση Στίβενσον για την εσωτερική αγορά. Να δώσω λοιπόν καταρχάς το λόγο στην κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες, απλά να πω ότι χθες είχαμε έναν τριμερή διάλογο, θα έχουμε και έναν σήμερα Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι κόκκινες ε, γραμμές. Έχω την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο καταβάλει προσπάθειες να κινηθεί προς τη δική μας κατεύθυνση και εμείς ε, το ίδιο προσπαθούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι η αποφασιστική συνεδρίαση θα είναι η αποψινή. Είμαι ε, αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα σήμερα ε, και μόνο για το λόγο ότι και οι δύο πλευρές δείχνουν σεβασμό απέναντι στην άλλη. Και στόχος μας ε, είναι να πετύχουμε μια μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά δεν θέλω να τις αναφέρω εδώ σήμερα, διότι νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις. Σήμερα πάντως φαίνεται ότι απόψε θα ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρωτούστ. Πριν ανοίξουμε τη συζήτηση για την πρόοδο σχετικά με τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ε, αναρωτιέμαι αν η Επιτροπή μου επιτρέπει να παρουσιάσω την έκθεσή μου, διότι πρέπει να πάω στην έκθεση ΑΦΕΤ για να συζητήσω ένα θέμα που έχει να κάνει ε, με το ΡΑΚ, ε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλίας. Ε, αν δεν έχει κανείς αντίρρηση θα ήθελα να το κάνω αυτό ε, χαίρομαι που τελικά πετύχαμε ε, συμφωνία όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγορά ε, κατά το τελευταίο τριμερή διάλογο. Έχουμε ακόμα μια τεχνική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε κάποιε εκκρεμότητε, κάποια μικρά ζητήματα, αλλά τα βασικά ζητήματα έχουν ολοκληρωθεί όλα. Όσον αφορά την επισήμανση, είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Κάθε προϊόν λοιπόν θα πρέπει να, επιτρέ... να περιέχει την επιστημονική ονομασία, τον ε, εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και την περιοχή όπου αλλιεύθηκε δεν θα πρέπει να ε, προκαλούν διακρίσεις ούτε να είναι παραπλανητικές οι επισημάνσεις. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία αλίας, η ημερομηνία εκφόρτωσης και άλλες ενδεχόμενες πληροφορίες αν θεωρούν ότι αυτό ε, θα τους δώσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η τελική γνωμοδότηση ζητάει από την Κομισιόν να υποβάλει έκθεση προς την Κομισιόν σχετικά ε, με τις ε, επισημάνσεις καθώς και με ε, μια ευρωπαϊκή οικολογική επισήμανση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα θα δώσει τέλος στο σύστημα των πολλών διαφόρων οικοσυστημάτων που έχουν προκαλέσει σύγχυση τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο θέμα είναι η κατεξοδότηση πράξης και οι εκτελεστικές πράξεις και χάρη στις ε, νομικές μας υπηρεσίες που υπέβαλαν ε, πρόταση κειμένου ε, συμφωνήσαμε για όλα τα επίμαχα σημεία. Πρέπει να φροντίσουμε οποιαδήποτε συμφωνία πετύχουμε να μην υπονομεύει την θέση μας απέναντι στο δικαστήριο και να προστατεύει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο δέχτηκε την ε, αναδιατύπωση μας ε, για τα άρθρα για τις οργανώσεις παραγωγών, ε, αλλά επίσης θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανιχνευσιμότητα των προϊόντων. Έτσι λοιπόν οι οργανώσεις παραγωγών θα προωθούν θα οργανώνουν συστήματα εκπαίδευσης για τα μέλη τους ε, και θα ε, συμβάλλουν στην ε, αύξηση της, επιλεξιμότητας, των, της επιλεκτικότητας των αλληλευτικών εργαλείων. Στόχος είναι σύγχρονος εξοπλισμός να χρησιμοποιείται προς όφελος του τομέα. Υπάρχουν παραδείγματα καλών αγορών που λειτουργούν με επιτυχία σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν ε, να ε, διευρύνουμε τη χρήση των ε, ηλεκτρονικών αγορών συνδέοντας τις με συστήματα VMS. Οι οργανώσεις παραγωγών έτσι θα μπορέσουν έτσι να βελτιώσουν τις αγορές για κάποια είδη, αποφεύγοντας τις ελλείψεις ή την υπερπαραγωγή. Θα χρειαστεί και βοήθεια από το Ταμείο Θαλάσσης και για να βελτιωθεί το σύστημα αυτά. Οποιαδήποτε βαρέλωση στην ελεύθερη αγορά όπως είναι το σύστημα απαγόρευση ή το σύστημα τιμών κίνησης είναι ε, θέματα που έπρεπε να χειριστούμε με πολύ προσοχή στον τριμερή διάλογο. Γνωρίζω ότι 45 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την ε, κατάψυξη ε, ηχθείων ε, σε περιπτώσεις όπου οι δαπάνες αποθήκευσης μπορούν να καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία, την Επιτροπή, την Ιρλανδία την Ιρλανδική Προεδρία και την ε, Κομισιόν για την ε, συνεργασία ε, και, την, και τις σκληρές προσπάθειές τους. Η πρώτη νομοθετική έκθεση ήταν αντικείμενο ευρείας συμφωνίας και ελπίζω και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στους τριμερείς διαλόγους για το βασικό κανονισμό. Θα ήθελα να ε, ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Ρόντοστε, σχετικά με τα αποτελέσματα του ε, τριμερούς διαλόγου και επίσης αν θέλει κανείς να σχολιάσει αυτά που μόλις είπα για τον ε, κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς. Θα δώσω πρώτο λόγο στην κυρία Καφία Τεπιέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να εκφράσω διαφωνία, αλλά υπάρχει κάποιο ε, θέμα σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση αγορά. Ε, ε, διάβασα στον τύπο ότι η συμφωνία ήταν με ομοφωνία. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Εγώ είμαι σκιώση ηγετρία για τους σοσιαλιστές και συμμετείχα επικοδομητικά σε όλες τις συνεδριάσεις. Έκανα προσπάθεια χρησιμοποιώντας και την νομική μου εμπειρία και σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία που μας βοήθησε πολύ. Αλλά αυτή η διαδικασία μου φάνηκε εμένα προσωπικά ε, υπερβολικά πιεστική από πλευράς χρόνου δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να μας υποβάλει ένα κείμενο μόλις 24 ώρες πριν και να πρέπει να το σχολιάσουμε σε τόσο στενές προθεσμίες. Πολύ δε περισσότερο που το κείμενο αυτό δεν είχε και μεγάλη σχέση με τις γενικές γραμμές που είχαμε εγκρίνει στην Ολομέλεια. Το ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, το άρθρο 42 ε, και την ετικετοθεσία ε, για, τις, ε, για τα αλλιεύματα της παράκτειας και εραστεχνικής και μικρής κλίμακος αλίας που πολλούνται 24 ώρες μετά την αλλιευσή τους ως νοπά. είχαμε ένα πρόβλημα με αυτό διότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτή τη μικρή κλίμακος αλία, την παράκτη αλία ιδιαίτερα ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης ε, έτσι ώστε να δουν αυτοί οι άνθρωποι ότι τους λαμβάνουμε υπόψη και δεν τους ε, αγνοούμε ε, η, η ανείχνευση η ανιχνευσιμότητα εξασφαλίζεται μέσω του, του barcode και μάλιστα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια ε, οπότε ε, είχαμε υποβάλει μια συγκεκριμένη τροπολογία την οποία, στην οποία επέμεινα για αυτό το λόγο. Και θέλω να πω το εξή, το Συμβούλιο εξ αρχής ε, ήταν αδιάλακτο. Δεν δέχτηκε ούτε, την ούτε για την ημερομηνία εκφόρτωσης που δεν χρησιμεύσε τίποτε. Την τροπολογία αυτή δεν δέχτηκε ούτε για την ημερομηνία εκφόρτωσης. Διότι αυτή είναι μια πληροφορία που έτσι κι δεν χρειάζεται. Επίσης ε, αρνήθηκε και την εθελοντική φύση. Την, ε, τη σήμανση αυτής. Ε, το κείμενο αυτό μπορεί πραγματικά να πλήξει θανάσιμα την αλία μικρής κλίμακας και την παρακτιαλία. Εκτός το ότι δεν ξέρουμε πότε, από πού και πώς στην τρίτη τελευταία συνεδρίαση της ε, διαπραγμάτευσης ε, ήρθε ένα mail το οποίο συμφωνώ, με το οποίο συμφωνώ. Μας λέγανε τι διαπραγματεύση είναι αυτή που εμείς υποχωρούμε σε όλα και το Συμβούλιο δέχεται τίποτα από εμά. Το, το μόνο που δέχτηκε το Συμβούλιο τελικά ήταν ορισμένα αλληλευτικά εργαλεία να προστεθούν στην ετικέτα. Σαν να ήταν αυτό αρκετό, σαν να αποτελούσε αυτός εγγύηση για τους ε, πολίτες μας που ε, θέλουν να καταναλώνουν ε, ψάρια από τη θάλασσα και όχι χθιοκαλλιέργειας ούτε ψάρια που έχουν μεγαλώσει με χθιάλευρα ή με πλεονάζοντα αλλιεύματα. Συνεπώς αν θέλουμε μέσω, του, μέσω κανονισμών να ε, προωθήσουμε ένα τμήμα του κλάδου με τα ποιητές για παράδειγμα ε, κρύβοντας πώς αλλιεύουν ή για να προστατεύσουμε ε, συγκεκριμένες σημαίες διότι δεν θα αναφέρονται δεν θα αναφέρεται η σημαία του σκάφους για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι κινέζικα σκάφη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά αλλιεύουν, μεταποιούν και πολλούν τα αλλιεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εκπροσωπούμε τους δικούς μας πολίτες και οι πολίτες είναι αυτοί ε, οι οποίοι πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας. Μιλάμε για, ένα, για μια Ευρώπη των πολιτών, δεν μιλούμε απλώς για ένα οικονομικό κλάδο. Αναγνωρίζω αφενός ότι ο κύριος Στίβενσον προσπάθησε να μας ενώσει, να μας εισπυρώσει κλπ. κλπ. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ε, δεν είχε τα, την επιτυχία ε, που θα ήθελε. Ε, εγώ θα υποστήριζα ένα κείμενο που δεν θα περιλάμβανε τουλάχιστον το άρθρο 42 όπως έχει. Γιατί ε, αν δεν δώσουμε τον ορισμό της ε, ασθενικής αλίας, αλίας μικρής κλίμακας, υπαράκτης αλίας κλπ, εντάξει. Ε, αν ε, δεν πούμε από πού ακριβώς προέρχεται το ψάρι, εντάξει, πάλι το δέχομαι. Αλλά αν επιπλέον ε, ε αλλά αν τελικά ε, δεν μπορούμε να περάσουμε τη γνώμη μας ούτε ε, στην ε, διάκριση ανάμεσα μεγάλων ελευτικών σκαφών και μικρών σκαφών αλληλείας μικρής κλίμακας, τότε ε, ποιος είναι ο ρόλος μας εδώ πέρα. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας θα έχουν πληροφορίες αρκετές έτσι ώστε να ξέρουν τι τρώνε. Έτσι κι αλλιώς αυτό ισχύει για τα άλλα τρόφιμα. Δεν είναι δυνατόν ε, από τη σήμανση της αλίας να λείπουν αυτές τις πληροφορίες. Και όταν μιλώ για τις ετικέτες δεν μιλώ για τον barcode, μιλώ για όλα αυτά που είδατε κι εσείς. Σε όλες τις ετικέτες, φωτογραφίες ετικετών, ε, στις ε, οποίες, είδατε κι εσείς και αναφέρετε το είδος με το εμπορικό του και το επιστημονικό του όνομα, ε, το, το μέρος από το οποίο αλλιεύτηκε κλπ δεν είναι δυνατόν από μια μεριά να κάνουμε εκστρατείε για να διδάξουμε στο κοινό να τρώει υγιεινά και από την άλλη μεριά να φέρουμε αυτές τις πληροφορίες από τη σήμα της. Πώς θα μπορούσα εγώ να συμφωνήσω. Δεν συμφωνώ. Και δεν υπάρχει και κανένα λόγο να βιαστούμε. Είμαστε σε πρώτη ανάγνωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μα βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό στην πρώτη ανάγνωση. Να συμφωνήσουμε, αλλά κάτι θα πρέπει, κάπου θα πρέπει να υποχωρήσει και το Συμβούλιο. Ή μήπω θα υποχωρήσει μόνο σε αυτά τα οποία ενδιαφέρουν ε, ένα συγκεκριμένο τμήμα ε, του κλάδου της ηχθειοκαλλιέργειας. Ε, επιμένω, η πλησιοφορία ήταν με πλειοψηφία. Η ομάδα των σοσιαλδημοκρατικών δεν υποστήριξε επουδενή σε καμία στιγμή αυτή την έκθεση. Ιδιαίτερα το άρθρο 42 που είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να απαιτήσουμε. Ευχαριστώ και λυπάμαι πολύ λυπάμαι βαθιά, που χρειάζεται να πω με τέτοιο ρητό και ομό τρόπο ε, την γνώμη μας. Η διαφορά μας όμως είναι τεράστια, μας χωρίζει ένα τεράστιο ε, χάσμα. Ε, ε, το Συμβούλιο έδειξε πραγματικά, δεν έδειξε καθόλου γενναιοδορία. Ευχαριστώ κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να περάσω στο βασικό κανονισμό και ξέρω ότι οι συνάδελφοι εδώ προετοιμάζονται για μια μακρά νύχτα και μάλιστα φαίνεστε ότι έχετε ήδη περάσει μια πολύ μεγάλη νύχτα. Ε, οι απορρίψεις καταρχάς, ξέρω ότι βρίσκεται πολύ ψηλά ε, στο θεματολόγιο του εισηγητή ο κανόνας δε είναι 5% όλων των αποθεμάτων. Ορισμένες φορές ε, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι προφανές και επομένως θα πρέπει ίσως να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ε, κάποια, ε, ε περιορισμός αλληλευτικό ταξίδι. σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξίζει τουλάχιστον τον κόπο περιορισμός και να είναι καλύτερος από ό,τι είναι τώρα. Δεύτερον, δεν το έχετε στο κατάλογο των θεμάτων που σας απασχολούν, δεν είναι στην προτεραιότητά σας ε, κυρία Συγήτρια, αλλά τα μεσοπρόθεσμα σχέδια κατά την άποψή μου είναι καλό το γεγονός ότι το Συμβούλιο θέλει να συστήσει μια νέα task force για να προσπαθήσει να λύσει τις δυσκολίες μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Από ό,τι φαίνεται οι Λιθουανοί κατά πάσα πιθανότητα θα το συνεχίσουν ε, το θέμα αυτό και θα προχωρήσει. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, μια δέσμευση ότι θα γίνει κάτι στο επόμενο τρίμηνο, θα γίνει μια πρώτη συνεδρίαση, διότι θα ήταν κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία και αυτό το θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ καιρό στην Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια και περνάει από τη μία προεδρία στην άλλη και την άλλη και την άλλη και το σέρνουμε πίσω μας, να τελειώσει. Και αν κατάλαβα καλά, εάν προκύψει θα συζητηθεί στο ε, τεχνική συνεδρίαση, όχι στις συνεδριάσεις που κάνετε εσείς για το τριμερή διάλογο. Μήπως θα μπορούσατε να μιλήσετε ιδιαίτερως με την Προεδρία και να τους πείτε μήπως θα μπορούσατε να μας καθορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για να δούμε όλοι και τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί είμαι σκιώδη εισηγήτρια στον ε, βασικό κανονισμό. Δεν χρειάζεται να σταθώ σε οτιδήποτε έχει ήδη συζητήσει η συγκήτρια, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για την κοινή οργάνωση αγοράς, ε, παρά το γεγονός ότι ε, συμφωνώ και εγώ με το πάθος της Λόλα για τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές. Δώσαμε όλη μάχη για να συμπεριλαμβάνονται όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και μάλιστα να είναι υποχρεωτικές τις ετικέτες. Δεν είμαι τόσο απασιόδοξη όσο και η Λόλα για το τι ακριβώς προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι ένα στοιχείο το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους καταναλωτές και επιτύχαμε είναι ότι θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή της περιοχής στην οποία αλλιεύεται το προϊόν και θα είναι και κατά τρόπον ώστε να είναι σαφές ε, στους καταναλωτές. Δεν θα γράφει πια ΦΑΟ 27, ΦΑΟ 46, θα πρέπει να λέει Βόρεια θάλασσα, θάλασσα της Ιρλανδίας, Βαλτική, θάλασσα, Κατεγάκης, ε, ε, κόλπος του Βισκαϊκού κλπ. κλπ. Ε, το, περιοχές δηλαδή που θα είναι κατανοητές στον καταναλωτή και θα υπάρχει ίσως και ένας χάρτης ή ε, μία εικονίτσα που θα δείχνει πού αλλιεύεται το προϊόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος και αυτό επετέχθη χάρη στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι λοιπόν γι' αυτό. Ένα άλλο ε, θέμα το οποίο πέρασε χάρη σε εμά είναι ότι οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αλλιεύεται το προϊόν ε, είναι και πάλι υποχρεωτικές. Θα γνωρίζουμε λοιπόν αν ε, ε, είναι παραγαδιάρικες, στράτες, είναι κλοβών, η αλλίευση, όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και αυτές είναι πληροφορίες που ο σύγχρονος καταναλωτής τις εκτιμά. Και το συμπεριλάβαμε και αυτό. Είναι αλήθεια ότι θυσιάσαμε πολλά πράγματα διότι το Κοινοβούλιο ήταν υπερφιλόδοξο, ε, θέλαμε να υπάρχει και το κράτος σημαίας ε, του σκάφους ε, που αλλιεύει τα ψάρια. Θέλαμε να ξέρουμε και πολλές άλλες λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά την ημέρα αλλιεύσης και την ημέρα εκφόρτωσης. Αυτά τα αρνήθηκαν όλα στο Συμβούλιο δυστυχώς. Νομίζω όμως και θα συμφωνήσει και η συγγήτρια νομίζω από αυτού ότι θα μπορούσαν ίσως να δίνονται και, και ο εισηγητής συγγνώμη ε, οι πληροφορίες αυτές οικειοθελώς από τους αλληλείς και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα το κάνουν. Ένα από τα θέματα τα οποία δεν ήταν επιτυχή ήταν ε, περαιτέρω πληροφορίες για τα μεταποιημένα προϊόντα. Αυτό ήταν προσωπική μου αποτυχία νομίζω, αλλά δεν ήταν στην επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ λοιπόν να κατηγορήσω τον εισηγητή που δεν κατάφερε να περάσει συγκεκριμένη πληροφορία. Ε, φταίει μάλλον η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που δεν υποστήριξε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πιστεύω ότι κάνατε καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λεβίν, ο κύριος Στίβενσον. Καταρχήν, να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Κρίστα Σήμερα είχαμε γεύμα με την Λιθουανική Προεδρία, με τον Υπουργό και συζητήθηκαν τα πολιετή σχέδια ως στοιχείο κλειδί της συζήτησης. Αυτός προσβλέπει σε, σε, σύντομη, σε, σε μια συνάντηση γρήγορα με την Task Force ε, και εγώ πρότεινα το Συμβούλιο να καλέσει τον πρόεδρό μας να τους ενημερώσει αυτοπροσώπως για το πρόβλημα. Του άρεσε η ιδέα και είπε ότι θα την ε, σκεφτεί. Έχουμε θέσει λοιπόν το θέμα στην κορυφή του θεματολογίου και γνώριζε πολύ καλά ότι αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα. σε απάντηση προς την κυρία Καρσία γιέρο Δολόρες. Εκτιμήσαμε τις ε, πολλές παρεμβάσεις σου στις πολύ ωραίες ε, ε, συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου. Θυμάμαι καμιά δύο περιπτώσεις όπου είχες ε, διαφορετική άποψη, αλλά σε δύο περιπτώσεις που είπες ότι ήθελες να σημειωθεί η αντίθεσή σου, την απέσυρες τελικά, κάτι που εκτιμήσαμε όλοι. Και γι' αυτό είπα ότι ήταν ομόφωνο το τελικό μας ε, αποτέλεσμα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ε, ήσουν αντίθετοι με κάποιο από αυτά τα σημεία και όταν μιλούσες για την προστασία των ε, συμφερόντων των ε, αλλιών μικρής κλίμακας. Το έχουμε κάνει αυτό. Έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα διότι μπορούν να προσφέρουν στο κοινό φρέσκα ψάρια που έχουν αλλιευτεί την ίδια μέρα. Δεν έχουν χρόνο ε, για επισημάνσεις, για barcodes και τέτοια. Συνήθως χρησιμοποιούν πίνακες, και είπαμε ότι αυτό μπορούν να το προωθήσουν σε εθελοντική βάση, αλλά υποχρεωτική ήταν η ημερομηνία λήξεως, η ημερομηνία ε, κατανάλωσης ε, κατά προτίμηση πριν να πω. Ε, σε ευχαριστούμε που συμφώνησες. Νομίζω ότι αν διαβάσεις προσεκτικά το τελικό αποτέλεσμα θα δεις ότι πολλοί από ε, τους φόβους σου ε, είναι αβάσιμη και μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα ωφελεί τον τομέα και ιδιαίτερα ε, τους αλληλείς μικρής κλίμακες. Όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο είχαμε εξετάσει. Το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου ε, εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση της έκθεσής μου, αλλά ε, ετοιμάζεται μια νέα έκθεση που θα καλύψει το θέμα αυτό. Κρίμα που συνεχίζουμε να επανερχόμαστε στο θέμα της επισήμανσης, ε, διότι έχουμε τόσους άλλους κανονισμούς που τελικά μπερδεύονται και οι καταναλωτές και ίδιοι η παραγωγοί. Πάντως το θέμα αυτό θα το χειριστούμε αλλού, όχι στη δική μου έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Εδώ Μιλάμε για τις ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αλληλεία ειδών βαθέων υδάτων ε, στον Βόρειο Ατλαντικό. Και ουσιαστικά μία προϋπόθεση υπάρχει. Α, αυτό είναι το επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη. Παρακαλώ θα μου δώσετε το λόγο στο επόμενο θέμα. Ζήτω συγγνώμη. <laughs> Η κυρία Ροντούστ. Θα ήθελα πολύ σύντομα να απαντήσω στον Chris Davis. Στον βασικό κανονισμό έχουμε τα πολιετή σχέδια ως σπονδυλική στήλη του βασικού κανονισμού. Και όπου είναι δυνατόν, ζητάμε από το Συμβούλιο επιτέλους να αναγνωρίσει την ε, συνθήκη της Εισαβόνα ε, και να μας πάρει σοβαρά. Ο Στρούαν αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, στους τριμμένους διαλόγους πιέσαμε πολύ, καταστήσαμε σαφές, επιμείναμε ε, τα πολιετή ε, προγράμματα να εφαρμοστούν και να, ε, και να αποφασίζουμε κι εμείς. Επίσης, όσον αφορά τις απορρίψεις, είπαμε ότι θέλουμε μηδενικές απορρίψεις, αλλά είπαμε ότι τελικά μπορούν να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις, διότι μας έπεισαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι απαραίτητο. Δεν συμφωνούμε όμως καθόλου με το θέμα των ποσοστών που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε εάν ε, αυτά θα έχουν να κάνουν με ε, τα είδη ή με τα αποθέματα. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα αλλιεύματα, αλλιώς, για συγκεκριμένα αποθέματα, αλλιώς δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος. σε εμπιστευτική συζήτηση με τον πρέσβη χθε το βράδυ. Του είπα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα απόψε. Αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να επιμείνουμε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Αγέρο. Κύριε Στίβενσον, εν συντομία, εξ αρχής αναγνώρισα και εξακολουθώ να αναγνωρίζω ότι εσείς κάνατε μια προσπάθεια και οι υπόλοιποι επίσης. Εμείς οι υπόλοιποι. Αυτή η προσπάθεια στις δύο πρώτες συναντήσεις κατέληξε μια συμφωνία ε, για λόγους συμβιβασμού και ε, άλλαξα θέση σε ορισμένα θέματα. Στην τρίτη όμως συνεδρία στις 8 Μαΐου από την οποία υπάρχει γραπτή η παρέμβαση μου την είχα στείλει από την προηγούμενη μέρα. Ε, σε αυτή την τρίτη συνεδρίαση ε, ανέφερα ποιε είναι οι πτυχέ στι οποίε δεν συμφωνούμε. Για παράδειγμα το 42-2 και το 42-1, τα δύο αυτά εδάφια. Για τα οποία είπα αυτή είναι η ε, συμφωνία της ε, Ολομέλειας, δεν είπα τίποτα παραπάνω και μάλιστα με υποστηρίζουν σε αυτό οι οργανώσεις των παραγωγών, οι οργανώσεις των αλλιέων κλπ. Το να είναι ε, υποχρεωτική η σήμανση ε, θα τους ε, βοηθούσε να δώσουν αξία στο προϊόν τους και έχουν χρόνο. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να, να καταστεί σαφές ότι στην τρίτη συνεδρία στις 8 Μαΐου και λυπάμαι γι' αυτό, έτσι, γιατί η κυρία Λεβίν ικανοποιήθηκε σε αυτό που ζητούσε ε, και γι' αυτό το λόγο συμφώνησε τελικά. Ε, λοιπόν, ε, δεν συνέβη το ίδιο με εμά. Εμεί είχαμε πει για την ημερομηνία αλίευση, είχαμε πει για τα αποκατεψυγμένα προϊόντα επίσης. Είχαμε υποβάλει μια τροπολογία, δύο σημαντικά πράγματα για τα, για τα οποία οι προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και να ανακοινωθεί ομοφωνία. Γι' αυτό το λόγο ήταν έκπληξη που διάβασα την επόμενη μέρα ε, στον τύπο ότι ε, εξασφαλίστηκε η ομοφωνία. Μπορεί να κάνω λάθος έτσι, αλλά η δική μου, προσωπική, η μου άποψη δεν είναι η προσωπική μου άποψη, είναι άποψη και πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των αλλιών κλπ. Αλλά αυτή είναι η άποψή μας. Ε, ασφαλώς και έχουμε χρόνο να συνδιαλλαγούμε και να συμφωνήσουμε το τελικό έγγραφο δεν βρίσκεται στα χέρια μας, τουλάχιστον όχι στα δικά μου. Συνεπώς δεν μπορώ να ερμηνεύσω κάτι που δεν έχω διαβάσει. Αν υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε διάλογο θα το κάνουμε. Γιατί ο στόχος είναι μια συμφωνία που να μην ε, απομακρύνεται από την πλειοψηφική απόφαση της Ολομέλειας και να είναι προς συμφέρον όλων μας και όλοι να θεωρούμε ότι είναι θετικό, θετική. Ωραία. Τελείωσε η συζήτηση, λέει ο πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, σημείο 15. Ειδική όρη όσον αφορά την αλία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοατλαντικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού 2347-2002. Γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει γίνει με αυτή την έκθεση. Η, πρόταση αυτή, ε, για την πρόταση αυτή ακολουθείται η διαδικασία συναπόφαση. Τον Οκτώβριο είχαμε δει την Κομισιόν να μα παρουσιάσει την έκθεσή τη. Μετά κάναμε μια ακρόαση με τέσσερα πάνελ και πάνω από οκτώ παρεμβαίνοντε. Το, το Μάρτιο αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να υποβάλει μια αξιολόγηση αντικτύπου πρόσθετη που να λαμβάνει υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και η Κομισιόν μπορεί να μας παρουσιάσει τη νέα αυτή αξιολόγηση πλέον. Θα της δώσουμε λοιπόν τον λόγο και κατόπιν θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρσένη που είναι εισηγητής και βέβαια στους ευρωβουλευτές που θέλουν να παρέμβουν. Κομμάτια της Κομισιόν. Sí, señor Candela. El señor Candela, perdón. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες διαφάνειες εδώ να σας δείξω. είναι μια πρώτη απάντηση ε, στο αίτημα της Επιτροπής σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θα δείτε τώρα για να κατανοήσετε τι ακριβώς ερευνούμε, με ποιες μεθόδους και σε ποιους τομείς εργασίας και να απαντήσω και σε τυχόν προκαταρκτικές ερωτήσεις. Όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ακόμα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε. Εδώ λοιπόν έχετε τους τομείς ε, στους οποίους ε, ε, ξεκινάμε τις εργασίες μας προς το παρόν προκειμένου να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες στο Κοινοβούλιο για να το βοηθήσουμε, να το συνδράμουμε, να το ενημερώνουμε ε, για προτάσεις μας. Θα αναφέρω αναλυτικά κάθε ένα από τα τρία σημεία, αλλά αυτοί είναι οι τρεις βασικοί τομείς. Ανάλυση του ε, GIS, του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, Κοιτάμε επίσης ε, τα πρόσφατα δεδομένα που διατίθενται μέσω του πλαισίου συλλογής δεδομένων και επίσης θα σας πω και λίγα πράγματα για τα βασικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε που είναι τα ουσιαστικά για τη συγκεκριμένη πρόταση. Ε, Επιτροπή Αλίας έθεσε μια συγκεκριμένη ερώτηση για, αυτό το συγκεκριμέ... για ένα από τα συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά πρέπει να τα αναφέρω όλα, θα δείτε εντός λίγο γιατί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο από τα τρία ζητήματα, το GIS, το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, εδώ προσπαθούμε ε, λίγο πολύ να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς ε, περιλαμβάνει αυτό το σύστημα και τι σκοπό έχουμε εμείς να κάνουμε με αυτό. Το GIS είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα και όχι μόνο στην Αλία αλλά και σε άλλους τομείς είναι μια τεχνολογία, ένα λογισμικό που βασίζεται ε, στη συγκεκριμένη τεχνολογία και συλλέγει ε, μεγάλο αριθμό δεδομένων σε γεωγραφικό πλαίσιο. Ουσιαστικά τα τοποθετεί στο χάρτη. Σε αυτή την περίπτωση ε, τι μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό το λογισμικό, να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων των σκαφών που συμμετέχουν στην αλληλεία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βάσει τις γεωγραφικές τους θέσεις και την γεωγραφική κίνηση τη δραστηριότητά τους. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος ε, και με τον όρο ποιος εννοώ ποιος αλλιέας ε, τι αλλιεύει, πότε, ε, τι ακριβώς και πόσα. Η πηγή μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι πηγές χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε δεδομένα από το VMS και από το μητρό του σκάφους, τα οποία παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Τις έχουμε ζητήσει αυτές τις πληροφορίες ήδη από πέρσι και κάθε πληροφορία που λαμβάνονται από το μητρό του σκάφου και οι θέσει που δίνονται μέσω του δορυφορικού συστήματο του VMS ε, και έχουν δηλώσει αλλιεύματα βενθοπελογικών ειδών και όταν λέω βενθοπελογικά είδη ε, αναφέρομαι στα είδη τα οποία αναφέρονται στην πρόταση. Όταν λέμε λοιπόν βενθοπελαγικά είδη αναφερόμαστε σε αυτά τα είδη. Ζητάμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη δεδομένα ε, από τρεις ε, πλήρεις χρονιές, από το 2009 μέχρι το 2011 και πρέπει να σας πω ότι απάντησαν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά δεν ε, μπορούσαν όλα τα κράτη-μέλη να μας δώσουν πλήρη στοιχεία για όλες τις χρονιές και στην πραγματικότητα έχουμε πλήρη στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη μόνο για το 2011. Επομένως, στην ανάλυση μας θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο για το συγκεκριμένο έτος. Ε, όποιο κράτος μέλος, έχει οποιοδήποτε σκάφος που έχει δηλώσει αλλιεύματα βενθοπελογικών ειδών, οποιασδήποτε ποσότητας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, μας έχουν δώσει τα στοιχεία. Έχουμε τα στοιχεία VMS λοιπόν για, όλες αυτές τις, ε, ε, για όλα αυτά τα ταξίδια και τα αντίστοιχα στοιχεία από το μητρό του σκάφους. Η ανάλυση είναι εν εξελίξη, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις πληροφορίες, θα σας δώσω συνοπτικά κάποιες πληροφορίες. Έχουμε 14 εκατομμύρια καταγραφές, όπως καταλαβαίνετε αυτές είναι πάρα πολλές. Τα στοιχεία που έχουμε από το Μητρό Σκάφους ε, ε, συνολικά είναι για 4.456 σκάφη, που σημαίνει ότι 4.456 σκάφη μας έχουν δώσει στοιχεία. Έχουν δοθεί λοιπόν εντός του 2011 στοιχεία για αλλιεύματα βενθοπελαγικών ειδών. Όπως γνωρίζετε αναφέρονται ανα κωδικό είδους και κάθε κωδικός είδους έχει ένα κωδικό τριών γραμμάτων και αν δείτε τα στοιχεία του μητρώου του σκάφους, αυτό που έχουν δουλάσει είναι ε, κωδικούς για 1116 διαφορετικά είδη. Αυτό σας δίνει μία εικόνα του πόσα πολλά διαφορετικά είδη αλλιεύονται σε αυτή την ε, περίπτωση και όχι μόνο τα μεθοπολογικά είδη. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κοινοποιούνται επίσης ε, ε, μέσω των μητρών, μέσω κωδικών και πάλι. Για το κάθε εργαλείο υπάρχει διαφορετικός κωδικός τριών γραμμάτων και πάλι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε 39 διαφορετικούς κωδικούς εργαλείων που είναι εντυπωσιακό αριθμό επίσης. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτά τα στοιχεία. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τα λιεύματα. Μπορούμε ε, μέσω αυτής της χαρτογράφησης να δούμε πως ε, οι άνθρωποι που αλλιεύουν ε, βενθοπελαγικά είδη ή ασχολούνται με βενθοπελαγικά είδη εν γέννη, αλλιεύουν αντίστοιχα στις ίδιες περιοχές με όλους τους υπόλοιπους στην πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα να επαληθεύσουμε ποιο ποσοστό αφορά τα αλλιεύματα βενθοπελαγικών ειδών ε, στη διάρκεια αυτών των ε, ε, ταξιδιών στη θάλασσα. Να σας υπενθυμίσω ότι αν ένα σκάφος ε, κάνει ένα αλλιευτικό ταξίδι και δεν αλλιεύσει καθόλου βενθοπελαγικά είδη, αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στο Μητρό. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονό ότι μπορούμε να κάνουμε και καταμερισμό αναείδο και μπορούμε να δούμε ποιε είναι οι βασικέ περιοχέ αλλή, ε, ε, ε, αλλιεύεται, παραδείγματος χάρη γρεναδιέρος του Ατλαντικού ή οποιοδήποτε άλλο, άλλο είδος και μπορούμε μετά να δούμε ε, με τι σκάφος αλλιεύονται, με παραγαδιάρικα, με γρηγρή, με οποιοδήποτε είδος σκαφών διαθέτουμε. Και αυτό φυσικά μας επιτρέπει στη συνέχεια να έχουμε μια βάση, να αναλύσουμε ε, κατά πόσον εξαρτώνται αυτοί οι άνθρωποι από τα συγκεκριμένα βενθοπολαγικά είδη βάσει των σκαφών που διαθέτουν. Μπορούμε επίσης να κάνουμε και ανάλυση ανακράτω σημαίας. Ε, τι γίνεται με τα σκάφη αυτά ένα σημαία που δίνει μια άλλη ενδιαφέρουσα οπτική γωνία για την οικονομική εξάρτηση που έχουν. Και αντίστοιχα μπορούμε, επειδή όλα αυτά τα σκάφη στα μητρώα που έχουμε ε, έχουν ένα λιμένα στον οποίο ανήκουν. Μπορούμε λοιπόν να συγκρατήσουμε τις δραστηριότητες και να τις ε, ε, καθορίσουμε με βάση το λιμένα και μπορούμε να έχουμε μια χαρτογράφηση όπου θα έχουμε όλα τα σκάφη που δηλώνουν ότι αλλιεύουν βενθοπελαγικά είδη, που επιστρέφουν, σε ποιο λιμάνι. Και έτσι γνωρίζουμε και την αξία των αλλιευμάτων και πόσα χρήματα φτάνουν στην κάθε περιοχή στο χάρτη. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο για ανάλυση ε, κόστους. Πολλά άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι οι βασικοί τομείς που σας ενδιαφέρουν. Κατόπιν έχουμε ένα άλλο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάση του υφιστάμενου πλαισίου συλλογή δεδομένων. Συλλέγονται δεδομένα για το σύνολο της δραστηριότητας και όχι μόνο για τα βενθοπελαγικά είδη. Και έχοντας τα δεδομένα για το σύνολο της δραστηριότητα, μπορεί να γίνει πραγματικά σύγκριση για να δούμε τι μερίδιο βενθυπολογικών ειδών έχουμε ε, για οποιοδήποτε τμήμα του στόλου σε σύγκριση με το σύνολο της δραστηριότητας και όχι μόνο ε, για τα αλληλεία μεθυπολογικών ειδών. η συλλογή δεδομένων, το πλαίσιο της συλλογής δεδομένων ναι, είναι ε, η πηγή από τις οποίες ε, τις, παίρνουμε πληροφορίες για τις δραστηριότητες ε, στους λιμένες και στις παράκτες περιοχές. Βλέπουμε για παράδειγμα πώς χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά ένα χαρακτηριστικό σκάφος σε ένα χαρακτηριστικό τομέα. Δεν έχουμε ατομικές πληροφορίες σε αυτό το σύνολο δεδομένων για κάθε σκάφος. Ε, δεν ξέρουμε αν το τάδε σκάφο απασχολεί 9 ή 10 ή 11 ανθρώπους, αλλά μέσω αυτού του συνόλου δεδομένων μπορεί να γίνει μια σύγκριση, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό σκάφο, για παράδειγμα μια τράτα ε, μήκους 18 ε, ε, και 24 για παράδειγμα και ξέρουμε ότι σε αυτή την περίπτωση συνήθως απασχολούνται χι άτομα και αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια προκειμένου να τα ε, διασταυρώσουμε με τα στοιχεία που έχουμε από το σύστημα GIS. Μπορούμε να διερευνήσουμε επίσης και κάποια στοιχεία για την ε, χοντρική προστιθέμενη αξία και επίσης το βασικό στοιχείο είναι το ποσοστό απασχολησιμότητας, δηλαδή ποσοστό που μπορούμε να έχουμε σε κάθε περιοχή απασχόλησης, ε, που σημαίνει ότι αυτό ανταποκρίνεται και στην οικονομία και το πόσο από αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στην αλληλεία βενθοπελαγικών ειδών. Θα θέλαμε πολύ ευχαριστώ να σας δώσουμε τα στοιχεία αυτής της ανάλυσης, τα αποτελέσματα, αλλά επειδή είναι τόσα πολλά τα στοιχεία δεν είναι έτοιμα τα ε, τα αποτελέσματα, αλλά θα είναι σύντομα έτοιμα και ελπίζω να μπορέσουμε να σας διανέμουμε τις πληροφορίες ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, σε δύο εβδομάδες το αργότερο. Να δούμε τώρα και λίγες διαφάνειες για θέματα που αφορούν στην έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχέση με τη διαχείριση των ε, αποθεμάτων βεβαιοπαλογικών ειδών. Τώρα, ποιες επιστημονικές γνώσεις πρέπει να έχουμε κατά νου ε, όταν συζητούμε αυτή την πρόταση, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει και ε, σημαντικά κονδύλια στην χρηματοδότηση αυτών των ε, τομέων έρευνας για να μπορέσουμε να αναλύσουμε ε, τα αποθέματα, την αλληλεία αυτών των ειδών ε, και τη διαχείριση και την παρακολούθηση. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε εδώ είναι ότι όταν εξετάζουμε τα επιστημονικά στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά να αναφερόμαστε σε στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Ε, αυτό ίσως θα το γνωρίζετε όλοι, αλλά μάλλον πρέπει να το επαναλάβουμε και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τα προγράμματα πλαίσιο, χρηματοδοτώντας διάφορα έργα. Τα έργα αυτά ε, εκτελούν τα καθήκοντά τους, κάνουν τις ερευνές τους και κατόπιν δημοσιεύονται άρθρα. Και αυτό ε, μεταφράζεται στην υλοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται για αυτά τα έργα. Ε, τα χρήματα ε, διατίθενται ακριβώς για δημοσιευμένα άρθρα τα οποία εξετάζονται και από τους ομολόγους τους. Ε, η επιστήμη, τα επιστημονικά στοιχεία έχουν αξία μόνο όταν λαμβάνουν και έγκριση από τους ομολόγους τους. Πρέπει λοιπόν όταν εξετάζουμε τα επιστημονικά στοιχεία να κοιτάζουμε και τι έχει δημοσιευθεί και αυτό είναι σημαντικό. Όσον αφορά λοιπόν το Deep Fishman, το Deep Fishman είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο ε, το έχουμε καθορίσει και στη σχετική βιβλιογραφία και τεκμηρίωση. Μας ενδιαφέρει η διαχείριση και η παρακολούθηση των ε, βενθοπελαγικών ειδών και αποθεμάτων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ε, έχει μια αξία της τάξης των 4 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. 3.765.139 ε, και η συνεισφορά του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3 εκατομμύρια περίπου. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 και περατώθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και αν δείτε τι δημοσιεύσεις έχουν προκύψει από εκεί έχουμε 7 τον αριθμό. Έχω βάλει και την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων Κόρντις ε, είναι μια ιστοσελίδα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί περιλαμβάνονται όλα τα ε, σχετικά άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν. Δεν έχω αντιγράψει τον κατάλογο βέβαια των άρθρων αυτών, μπορείτε κάλλιστα να τα δείτε στην ιστοσελίδα, αλλά στόχο έχουν ε, γνώσεις και επιστημονικά στοιχεία για καλύτερη αξιολόγηση ε, των ειδών. Έχουν εξετάσει διάφορα είδη και υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο ε, στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που δίθονται από τους ενδιαφερομένους για να βελτιωθούν τα αποθέματα και να βελτιωθούν και οι γνωμοδοτήσεις κάθε χρόνο για το τι ποσόστος θα πρέπει να αναλυεύεται κάθε χρόνο. Ε, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι εκεί επικεντρωνόμαστε. Αυτό είναι το στοιχείο που απασχολεί το πρόγραμμα Deep Fishman, καλύτερη γνώση των πενθαπελαγικών αποθεμάτων. Κατόπιν έχουμε δύο προγράμματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε εδώ. Και εδώ έχουμε την, άλλη πτυχή. Πού ε, γίνεται η αλληλεία και πώς επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Το Ερμιόνι είναι το μεγαλύτερο από τα δύο προγράμματα. Είναι εντυπωσιακό το ποσό που δίνεται, περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Ε, σχεδόν τα 8 εκατομμύρια δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε 202 δημοσιεύσεις. Οι ε, όσες αυτές δύο δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν πάρα πολλά στοιχεία για το ε, θαλάσσιο περιβάλλον, ε, τι αποτελέσματα έχουν, ε, τι γίνεται με τη βιολογία και τα οικοσυστήματα και πώς θα πρέπει να περιγράψουμε το ρόλο τους και Υπάρχουν και αρκετά άρθρα τα οποία είναι ειδικά αφιερωμένα στην ανάλυση των επιπτώσεων της αλίας για το συγκεκριμένο θαλάσσιο περιβάλλον. Εάν λοιπόν κάποιος μπορέσει να λάβει περισσότερες γνώσεις για το πώς λειτουργούν αυτά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, πόσο ευάλωτα ε, είναι ή δεν είναι και πόσο ε, συχνά εμφανίζονται στα δικά μας τα ύδατα και ούτω καθεξής, μπορεί στη συνέχεια κάποιος να αναλύσει λίγο καλύτερα τις συνέπειες της αλληλείας αυτών των ειδών. Αποτελεί προϋπόθεση. Ε, βεβαίως ε, δεν ασχολείται μόνο με την αλληλεία, ασχολείται με και τις συνέπειες που έχουν και τα υπόλοιπα στοιχεία. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα ε, στοιχεία, βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην αλληλεία βαθέων υδάτων. Όταν θα δείτε και την κατάλληλη έκθεση για όλα αυτά τα θέματα, θα κάνουμε και τον κόπο να σας παρουσιάσουμε όλες αυτές τις μελέτες που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Εδώ και πάλι έχετε και την ιστοσελίδα που μπορείτε να δείτε όλο τον κατάλογο των δημοσιεύσεων. Και τέλος μια τελευταία μελέτη, η Coral Fish. Η Coral Fish ε, αφορά το ε, θαλάσσιο περιβάλλον για τα, και τα βενθοπελαγικά είδη. Προσπαθούμε να ε, συγκεράσουμε εδώ τα καλύτερα στοιχεία των άλλων δύο τομέων στους οποίους επικεντρωθήκαμε σε άλλες μελέτες. Πρόκειται και για, σε αυτή την περίπτωση για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Η χρηματοδότησή του είναι αντίστοιχη με το Ερμιόνι, περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 6,5 διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις ολοκληρώθηκε και ε, μέχρι τώρα είχαμε 11 δημοσιεύσεις. Εδώ ασχολούμαστε με τα κοράλια ε, τα βενθοπελαγικά, ε, εξετάζουμε την βιολογία τους, ε, το πού βρίσκονται, τη δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων για να μελετήσουμε με κάποια ακρίβεια πού θα μπορούσαμε να έχουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά μοντέλα και υπάρχει και μια συγκεκριμένη μελέτη, μελέτη την οποία θεώρησα ότι είναι σημαντική σε ένα από αυτά τα 11 άνθρα έχουμε εάν ε, μια εξέταση του κατά πόσον αυτό το διαβόητο move on rule που ο κανόνας αυτός που φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι είναι αποτελεσματικός και προτείνονται κάποιες λύσεις για το πώς μπορεί να διατηρηθεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Μπορείτε να τα εξετάσετε όλα αυτά, έχουμε και τη σχετική στο σελίδα. Αυτό κάνουμε λοιπόν και αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να αναμένετε πολύ σύντομα θα ήθελα να ζητήσω και πάλι την υπομονή σας. Θα θέλαμε πάρα πολύ σήμερα να σας παρουσιάσουμε τα συνολικά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως επειδή ήταν τόσο μεγάλη η μελέτη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι τόσο καλό για το χρονοδιάγραμμά μας, αλλά είναι καλό από πλευράς ανάλυσης. Ε, αξίζει λοιπόν να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε να σας παρουσιάσουμε πληροφορίες που είμαι βέβαιη ότι θα θεωρήσετε ότι ε, θα σας διαφωτίσουν πολύ καλύτερα στη συζήτησή σας. Ε, είμαι στη διάθεσή σας τώρα κύριε Πρόεδρε για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Αρσένη. Πριν λάβουν το λόγο κατόπιν και οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αλλαγή στάσης των κρατών μελών, τα οποία τελικά δίνουν στοιχεία στην Επιτροπή και την ικανοποίησή μου γιατί η Κομισιόν μπορεί πλέον να μας δώσει απαντήσεις για όλα τα θέματα που ανησυχούσαν το Κοινοβούλιο. Πολύ καλή συνεργασία και πολύ, καλή, πολύ καλός σεβασμός ε, της θέσης του κάθε οργάνου στην νομοθετική διαδικασία. Περιμένουμε με ανυπομονησία το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή και όλοι οι παρόντες συνάδελφοι θα συμφωνούν ότι είναι πολύ ικανοποιητικό το επίπεδο ε, η ποιότητα μάλλον ε, της, το, αποτελέσματος που θα πετύχουμε με αυτά τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ε, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ικανοποιημένοι για την, από την βάση της νέας ε, αξιολόγησης. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω με αυτή την ευκαιρία αυτό που έχω πει επανειλημμένο στο παρελθόν, ότι αυτή η νομοθεσία έχει ως ε, στόχο πλευράς ε, Κοινοβουλίου να εντοπίσει ακριβώς τις ε, πολιτικές και τα εργαλεία για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για τα προβλήματα και τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης των, της αλλιάς βαθαίων υδάτων. Οπότε τα μέτρα που θα πάρουμε θέλουμε να είναι αναλογικά και εστιασμένα στα προβλήματα. Στόχος είναι να βρούμε λύσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφύγουμε να επηρεαστεί αρνητικά ο οποιοδήποτε άλλος τύπος αλίας. Γιατί ο στόχος μας είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα, όχι να δημιουργήσουμε άλλα. Θέλω να είμαι σαφής αυτό. Από την ε, δική μου πλευρά, αυτό το θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα, η έκβαση αυτής της μακράς διαδικασίας συζήτησης, διαλόγου, προσπάθειας να βρούμε μια συνένεση στην Επιτροπή μετά την υποβολή τροπολογιών. Μιλούμε για ένα ολόκληρο μήνα ε, προετοιμασίας των συμβαστικών προτάσεων προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ενιαία, σε μια τοποθέτηση. Συγχαρητήρια μια ακόμα φορά για αυτά που μας είπατε και περιμένουμε και τα αποτελέσματα για να τα χρησιμοποιήσουμε στις εργασίες μας. Merci, Ευχαριστώ, Κριτών, λέει ο Πρόεδρος. Ο λόγος του κύριου Άγνιου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα έχουμε πάρει λάθος τα πράγματα. Ανάποδα. Γίνονται σημαντικές παραβιάσεις στα βαθιά ύδατα. Φανταστείτε μια τάξη σχολική, όπου ο δάσκαλος ε, είναι ύποπτος για βιασμό. Ε, τι τι γίνεται. Ε, τον, τον ανακαλούν μέχρι ότου να στέλνουν την, τα καθήκοντά του μέχρι, να, μέχρι ότου να εκδικαστεί η υπόθεση. Τι γίνεται τώρα, αντί να κάνουμε αυτό στον βορειοανατολικό Ατλαντικό η Κομισιόν ρίχνει ακόμα περισσότερα χρήματα, ε, περνάνε τα χρόνια, ενώ όσο η αλία συνεχίζεται. Η Κομισιόν μας είχε ζητήσει ε, υπομονή. Εγώ πιστεύω ότι ε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Οι περισσότεροι από εμάς εκπροσωπούμε πολίτες ε, Μάλλον πολλοί από του ευρωβουλευτέ θέλουν την ε, καθυστέρηση γιατί εκπροσωπούν πολίτε που του ζητούν να συνεχίσουν να αλλιεύουν και μάλιστα μεγαλύτερε ποσότητε και του λένε γι' αυτό σα εκλέγουμε. Ε, ο αλλιευτικό στόλο του Ηνωμένου Βασιλείου πλήττεται. Και οι φορολογούμενοι ταυτόχρονα ε, με λύπη τους βλέπουν ότι χρηματοδοτούμε, επιδοτούμε ε, ξένους αλλιευτικούς στόλους που αλλιεύουν εκεί, στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, ενώ οι δικοί μας χάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Merci Monsieur Agnew. vous, Comme d'habitude, vous avez fait dans la dentelle. Donc, euh... Όπως ε, συνήθως κύριε Άγνιος, ήσασταν πολύ εύγλωτος. Chris Davis έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω μπερδευτεί. Τι ακριβώς ζητάει η Επιτροπή. Μας προτείνει. Μάλλον ε, θεωρεί ότι με τη δουλειά αυτή που μας έχει δώσει πολλές πληροφορίες θα πρέπει να αναστείλουμε την διαμόρφωση της νομοθεσίας αυτής μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα και ότι αν δεν έχουμε τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα. Πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα αυτά. Πρέπει να γνωρίζουμε και η Επιτροπή πότε θα μπορέσει να μα δώσει τι πληροφορίε αυτέ Μιλάμε για χρόνια ή μιλάμε για εβδομάδες. Και τώρα που έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Συναντήθηκα με ιδιοκτήτε αλλιευτικών σκαφών χθε. που αλλιεύουν στον Βορειοανατολικό ωκεανό, Ατλαντικό ωκεανό και λένε ότι ευχαρίστω να υιοθετήσουμε τις αρχές εδώ, ώστε να έχουμε βιώσιμη αλληλεία και να μην βλάπτουμε το οικοσύστημα κλπ. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τον τομέα της, αλλη... της αλληλείας και όχι εναντίον του. Πολύ ευχαρίστω θα ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις εάν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να πάρει τη μορφή νομοθετική τροπολογία, ώστε να εφαρμόσουμε με πρακτικό τρόπο την νομοθεσία. Το θέμα όμω είναι εάν θα μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους κείμενα. Αν μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα πρέπει να τα προσέξουμε πολύ προσεκτικά και ελπίζω ο εισηγητής ε, να εξετάσει προσεκτικά τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. θεωρητικό θα πρέπει να πάρω τώρα το λόγο, αλλά επειδή προεδρεύω θα το αφήσω για αργότερα. Ο λόγο στην κυρία Λεβίν, όχι, δεν έχει δει το λόγο. Νόμιζα ότι είχε σηκώσει το χέρι σου. Ωραία. Κάρμεν Φράγα. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη, ήμουνα σε άλλη συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Μου είπαν συνοπτικά τι μου περίγραψαν τι είπε, η μεθοδολογία που παρουσίασε είναι πολύ πιο πλήρης από αυτήν που ακολουθήθηκε στην προηγούμενη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου. Το Κοινοβούλιο δικαιολογημένα αποδεικνύεται ζήτησε επικαιροποίηση της προηγούμενης μελέτης, διότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη όλα τα κριτήρια, όλες οι συνιστώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κοινωνικο τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Η Κομισιόν βέβαια ακόμα επεξεργάζεται τα στοιχεία, αλλά έχοντας έρθει σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη και του, τους ε, κλάδους που επηρεάζονται, ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λίγα σκάφη στα οποία αναφέρθηκε η Κομισιόν χωρίς να δώσει συγκεκριμένο νούμερο και που θα επηρεαστούν από την πρόταση δεν είναι και τόσο λίγα τελικά. Έχω στοιχεία τη Γαλλία του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ισπανία, οπότε αυτά τα λίγα πλοία είναι πολύ περισσότερα, αυτά τα λίγα σκάφη, ε, οπότε η μελέτη αυτή θα είναι πολύ σημαντική. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξή. Αφού η Κομισιόν κάνει αυτή την αξιολόγηση και σε συνάντηση με τα αποτελέσματα ε, προτίθεται να τροποποιήσει την δική της πρόταση. Γιατί εδώ έχουμε μια καινούργια ανάλυση, μια καινούργια μεθοδολογία, ίσως τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν προβλεφθεί στην αρχή. Αν λοιπόν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν αυτό που κάποιοι από εμά πίστευαν, η Κομισιόν ε, είναι πρόθυμη να τροποποιήσει την πρότασή της. Δεύτερον, και έχω μιλήσει γι' αυτό με τον εισηγητή. Υπάρχει κάτι το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Κανείς δεν θέλει να υποστηρίξει κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Το πρόβλημα είναι η το κατά πόσον η εστίαση της Κομισιόν είναι σωστή. Γιατί πολύ ωραία όλα αυτά για τις παραβιάσεις κλπ. Αλλά αν όλοι θέλουμε τη βιωσιμότητα που όλοι τη θέλουμε και όλοι θέλουμε αυτός ο τομέας να διατηρηθεί, να επιβιώσει. Όμως από το 2002 που υπέβαλε την πρώτη πρότασή της η Κομισιόν ε, επήλθε μείωση 30% στην αλληλευτική προσπάθεια και ορισμένα από τα αποθέματα τα οποία πιο πολύ ε, αλλιεύουν οι ευρωπαϊκοί στόλοι έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακτηθεί και αυτό το είπαμε και σήμερα το πρωί. Συνεπώς τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αλλά όχι αρκετά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε λοιπόν. Ορισμένοι πιστεύουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ακραία και δεν θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί ένας λόγος είναι επειδή θα συνεχίσουν να αλλιεύουν άλλοι, άλλα σκάφη δεν θα είναι ευρωπαϊκά. Και τι θα γίνει τελικά, θα εισάγουμε τα δικά τους προϊόντα. Γιατί αυτή η απαγόρευση θα αφορά μόνο τους ευρωπαϊκού, τον ευρωπαϊκό στόλο. Συνεπώς, ο ΦΑΟ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι έχουν κανόνες που ενδεχομένως είναι πιο αποτελεσματικοί. Συνεπώς, περιμένω σύντομα τα αποτελέσματα και από τη βάση αυτών ίσως καταφέρουμε να βρούμε ποια είναι η πιο σωστή λύση και για τα αποθέματα αλλά και για τον αλλιευτικό μας κλάδο που ε, δρά, ε, δραστηριοποιείται επί ενός ανανεώσιμου, ανανεώσιμου, στόχου Ευχαριστώ κύριο Σκαντέκ Ε, καταρχάς και εγώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας εξηγήσατε λίγο τη μέθοδο εργασίας σας ε, για την αναθεώρηση των, ε, της μελέτης Ε, περιμένουμε με ανυπομονωσία την έκθεση. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις για τη μελλοντική αναθεώρηση της ε, μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασίζεστε σε γνωστούς ε, στόλους, ε, σκάφη που αλλιεύουν βενθοπολογικά είδη για να αξιολογήσετε ποια προτείνετε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Θα μου απαντήσετε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί κατά πάσα πιθανότητα θα έχει σωστέ εκτιμήσεις. Είναι λίγες οι πιθανότητες να μην είναι σωστές εκτιμήσεις. Ε, και γιατί λέτε ε, ότι θα μπορέσετε να στοχεύσετε σε σκάφη τα οποία ε, αλλιεύουν ε, ε βενθοπελαγικά είδη. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη ε, αλλιεύουν ε, συγκεκριμένα είδη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ανώτερες οι ποσότητες όταν είναι 100 κιλά τη φορά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση απορρίπτονται αυτά διότι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να προσμετρούνται στο συνολικό αλλιεύμα. Υπάρχει όμως τώρα η υποχρέωση εκφόρτωσης και αναγνώριση ως ε, βενθοπελαγική αλληλεία. Και εμείς θεωρούμε βενθοπελαγική αλληλεία, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ποσότητες άνω των 100 κιλών ανά ε, ταξίδι. Όλα τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιεύουν για λόγους επιβίωσης. Αν όχι όλα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έστω ότι έχουμε μία τράτα 25 μέτρων, που αλλιεύει καραβίδες σε 100 μέτρα βάθους ή σταματάει στα 500 μέτρα συγγνώμη, βάθους. Συνειδητοποιεί ότι ε, συγγνώμη, κάνει 4 με 5 ταξίδια την ημέρα και αλλιεύει ε, συγκεκριμένα κιλά την ημέρα θα ε, αλλιεύσει σε αυτή την περίπτωση 100 κιλό, ε, κιλά και αυτά δεν θα θεωρούνται όμως σκάφη τα οποία αλλιεύουν βενθοπολαγικά είδη, διότι δεν ξεπερνούν το ε, συνολικό αριθμό που, που επιτρέπεται. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τους απαγορεύσουμε την πρόσβαση στις ζώνες στις οποίες αλλιεύουν παραδοσιακά γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν ότι αλλιεύουν πάνω από 100 κιλό τη φορά δηλαδή θα πρέπει να πάρουν άδεια και δεν θα μπορούν για να συνεχίσουν να αλλιεύουν εκεί που αλλίευαν προηγουμένως. Επίσης λέτε τι μεθοδολογία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε σε αυτό προηγουμένως. Ε, στην ανάλυση επιπτώσεων ε, ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε αν θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που θα έχουμε από τις απορρίψεις ε, στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση το CSTIP e ή θα αναλύσετε όλα τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν ε, ε, αλία βενθοπολογικών υδάτων ή μέχρι κάποιο βάθος και αν μπορεί να γίνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, μας μιλήσατε για το Deep Fishman το πρόγραμμα αυτό ένα σκάφος θα μπορούσε να έχει και παρεπίπτοντα αλλιεύματα βενθαπολογικών ειδών, αυτή τη στιγμή αλλιεύει άνω των 100 μέτρων βάθος. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα μπορούσε να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνει πέραν των συστάσεων που κάνει η ΝΑΦΚ που προτείνει να σταματήσει σταδιακά αυτή η δυνατότητα. Ελπίζω ότι αυτή η επανεξέταση της μελέτης επιπτώσεων θα μας αναλώσει ακριβώς πώς έχει η κατάσταση, γιατί είναι τόσο κακή η κατάσταση αυτή τη στιγμή και θα μας δώσετε και τα στοιχεία τα οποία θεωρείτε εσείς ότι είναι σημαντικά. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και αυτά ήταν απλώς κάποια ερωτηματικά, αλλά πραγματικά αναμένουμε πάρα πολλά από αυτή τη μελέτη επιπτώσεων, διότι πρέπει να έχουμε και εικόνα, όπως είπε και ο Κρήτον προηγουμένως. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Euh, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σήμερα δεν θα ξαναρχίσουμε εις βάθος συζήτηση επί του θέματος. Ε, εμείς μεταξύ μας θα τη συνεχίσουμε με το καλύτερο πνεύμα ε, συνεργασίας, όπως προτείνει ο εισηγητής μας. Εγώ δεν θα ήθελα να προδικάσω, όπως κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, τα αποτελέσματα αυτής της ε, έρευνας και της μελέτης ε, που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι μία αναθεώρηση εις βάθος ε, όλων των στοιχείων που διαθέτουμε μέχρι τούδε. Τώρα, το κατά πόσον τα αποτελέσματα εκφύσεως ε, θα είναι διαφορετικά ή όχι, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, θα το δούμε. Και αυτό το οποίο αντιλήφθηκα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτά τα στοιχεία ε, από τα οποία λαμβάνεται περαιτέρω πληροφορίε, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε τι εργασίε μα. Αυτέ λοιπόν ε, οι περαιτέρω λεπτομέρειε θα μα δοθούν πολύ σύντομα. Είπατε ότι είναι σχεδόν έτοιμα. Ε, δεν είπατε αυτό στα αγγλικά βέβαια, αλλά στα, αγγλικά αυτό, στα γαλλικά αυτό μεταφράζω. Ε, ίσως και στην επόμενη φορά που θα είστε εδώ να σας ακούσουμε ή λίγο αργότερα, τέλος πάντων ε, σύντομα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια απόφαση. δεν χρειάζεται να ε, καθυστερούμε άλλο τις ε, κινήσεις μας. Έχει φτάσει κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε αφού θα έχουμε λάβει τις περισσότερες πληροφορίες και δεν θα ξεκινήσει τώρα μία στρατηγική ε, εξάντληση του ζητήματος. Πρέπει κάπου να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν αν θέλουμε πραγματικά αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα από πλευράς ε, βενθοπελαγικής αλίας να ε, βελτιωθεί και να, να μειωθεί το πρόβλημα και να πλαισιωθεί καλύτερα. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Α, συγγνώμη, κυρία Γκαρθία Ιέρο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις κάποιων ειδικών που εξέτασαν αυτή τη μελέτη. Είναι ακόμα πολύ αμφίσιμο το πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή δεν δίνει στοιχεία για το ε, ποιες χώρες αφορούν ποιους ε, στόλους και λέμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα για το στόλο, αλλά να βελτιώσουμε τα λιευτικά εργαλεία για να είναι καλύτερη αλία. Αυτό όμως θα πρέπει να ε, να το δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει σε τι στόλο αναφέρονται, με τι εργαλεία αλλιεύουν, σε ποιες περιοχές και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των χωρών μελών είναι αλληλένδετα, διότι υπάρχει μια περίπτωση στην οποία εξετάζουμε και τη δυνατότητα απαγόρευσης ε, και στην ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, συζητάμε και το θέμα να έχουμε προγράμματα διαχείρισης για να μην ε, ε, ξεπερνούμε τα όρια. Δεν μιλάμε για απαγορεύσει αυτέ καθ' αυτέ. Ε, θέλουμε να βελτιωθεί ο στόλο, να βελτιωθούν τα λεφτικά εργαλεία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αλίευση σε κάποιε περιοχέ, για παράδειγμα, όπω στην Αστούρια, όπου δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλα σκάφη, δεν έχουν πολύ ισχυρά εργαλεία. Και εκεί τους επιβάλλεται να αλλιεύουν κάποια συγκεκριμένα είδη τα οποία, ε, να μην αλλιεύουν συγγνώμη κάποια είδη τα οποία θα απαγορευτούν στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποια είδη τα οποία φτάνουν στις αγορές και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για κράτη σημαία ε, που μπορεί να μην είναι από την Κίνα αλλά ε, προφανώς ε, από πίσω είναι η Κίνα. Ε, και είναι πιο αδύναμες οικονομίες ε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε κάποιες χώρες που πρέπει να καταναλώνουν ε, ψάρια και δεν έχουν πρόσβαση εντός εισαγωγικών σε καλύτερης ποιότητας ψάρια. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, γιατί στη συνέχεια θα έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά προς το παρόν θα έπρεπε να καθορίσουμε τι είναι θεμελιώδες. Για να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση σαν αυτή που θα δημιουργήσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα στους συγκεκριμένους τόλους. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Αναφερόμαστε σε παραβιάσεις. Είναι πολύ ισχυρός αυτός ο όρος. Ε, μπορούμε να πούμε αν παραβιάζεται η νομοθεσία ή παραβιάζονται οι κοινοτικοί κανόνες, αλλά μηχανισμοί εποπτείας, μηχανισμοί παρακολούθησης, κυρώσεις, ε, είναι κατάλληλα αυτά, ε, έχουν αποτελέσματα, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο στόχος. Ε, μήπως ορισμένες φορές απλώς καθορίζουμε στο στόχο και μετά κάποιες χώρες τα τηρούν και κάποιες άλλες όχι. Ε, εγώ να σας πω τι βλέπω επιτόπου. Η χώρα μου είναι μία από αυτές τις χώρες ε, που είναι ε, πάρα πολύ αυστηρή όταν γίνονται εκφορτώσεις, βλέπει τι γίνεται, βλέπει τι συνέπειες υπάρχουν, είτε πρόκειται για αλληλεία ή αλληλευτικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε τα είδη που ε, είναι σε κίνδυνο σε βαθαία ύδατα ε, να μπορέσουν να προστατευτούν και να μην τα χώσουμε όλα στο ίδιο καζάνι και να μην αρχίσουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όλα τα βενθαπελαγικά είδη κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν ε, να μπουν στο ίδιο καζάνι και να υπάρχουν και κάποια είδη τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τη δέουσα ισορροπία είναι αμφίσιμο το κείμενο, ε, ελπίζω να υπάρξει πρόοδος με την έκθεση αυτή και θα πρέπει να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι καλό εφαλτήριο ε, αυτή η έκθεση και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο συνάδελφος Αρσένης ε, έχει κοινή λογική και μπορεί να συμπεριλάβει τα σωστά στοιχεία ώστε να έχουμε μια καλή έκθεση στο τέλος. Η Κομισιόν θέλει να παρέμβει. Κύριε Πρόεδρε, μου τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω τα σημεία που αποτελέσαν αντικείμενα ε, ερώτησης. Ε, να ξεκινήσω από τον κύριο Καντέκ, διότι αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστούν στη συζήτηση αυτή. Καταρχήν, σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου ότι εδώ συζητάμε όχι την απαγόρευση της αλίας μετράτα. καταργούμε βαθμιαία κάποιες ε, άδειες για αλία βαθέων υδάτων. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ο καθένας σήμερα έχει άδεια για αλία βαθαίων υδάτων, διότι αν δεν την έχει κανείς, τότε μόλις πιάσει κανείς παραπάνω από 100 κιλά σε οποιαδήποτε ε, ε, ε, μέρα δεν μπορεί να τα εκφορτώσει και θα πρέπει να τα πετάξει, να τα απορρίψει. Μπορεί λοιπόν να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν άδεια, θα πρέπει να απορρίψουν λοιπόν 100 κιλά ηχθείων και δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία. ο τρόπος που καταχωρούνται οι απορρίψεις ε, στα ημερολόγια των πλοίων ε, δείχνει μάλλον ότι το ημερολόγιο δεν επιτρέπει την καταχώρηση ε, αυτής της αλληλείας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι ε, ε, στο πλοίο που κάνουν υπολογισμούς σχετικά με τον κανονικό ρυθμό απορρίψεων και βγάζουν εκείνη τα στοιχεία, αλλά 100 κιλά είναι πολύ λίγο. Έτσι λοιπόν ένας αλληλείας θα πει είτε ότι αν δεν με ενδιαφέρουν τα ίδια αυτά, αν πιάσω 100 κιλά θα τα απορρίψω ή θα πάει κανείς ε, στο Υπουργείο του, θα ζητήσει άδεια και θα του δοθεί η άδεια. Ο Αλίες αυτός λοιπόν έχει μια τέτοια άδεια. Προφανώς θα έχει μία για ε, νότιο εγκλεφίνο, μία για τον ε, βόρειο εγκλεφίνο, μία για τα πλατήψαρα. τα χρειάζονται λοιπόν οι αλλοί τις άδειες αυτές. Κυρίες και κύριοι, σαφές εδώ είναι σίγουρο το ότι κανένας ε, δεν έχει ε, σύνθεση ε, των αλλιευμάτων του 100% από τη βαθιά θάλασσα. Η αλία βαθαίων υδάτων παραμένει κάτω από το 1% της συνολικής αλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που στοχεύουν στην αλία βαθαίων υδάτων και πάρα πολλοί αλλιεύουν τα ίδια αυτά ω ε, τα αλλιεύματα. Στόχος λοιπόν εδώ είναι να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τις ε, λεπτομέρειες αυτές, αλλά η Γενική Αρχή παραμένει. Η αλία βαθέων υδάτων παραμένει ε, ένα πάρα πολύ σκοτεινό μέρος της οικονομίας της αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε στη μελέτη αντικτύπου ότι ναι, αναγνωρίζουμε ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ε, τοπικά πολύ σημαντικές, ότι υπάρχουν ε, περιοχές ε, όπου διεξάγονται κάποιες επιχειρήσεις και πρέπει να σκεφτεί κανείς τι πρέπει να γίνει με τις περιοχές αυτές. Στην μελέτη αντικτύπου σας παραπέμπω πάλι στο θέμα του γαλλικού στόλου, διότι είναι ο μόνος που εξειδικεύεται που ειδικεύεται στην ε, αλία βαθαίων υδάτων ε, και πάλι το ποσοστό των ε, αλλιευμάτων βαθέων υδάτων είναι 40% σε σύγκριση με το 60% που είναι άλλα αλιεύματα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι το θέμα δεν είναι να απαγορεύσουμε τις στράτες, είναι να καταργήσουμε βαθμιαία άδειε οι οποίες καλύπτουν ένα σχετικά μικρό κομμάτι της δραστηριότητας των ανθρώπων αυτών. Σε θα μπορέσουμε εμείς να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα ανατομέα, αναπεριοχή κλπ. Αλλά η γενική εικόνα παραμένει ε, ε απαράλλαχτη. Γι' αυτό η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο ότι στις οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να ε, εξισορροπήσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Και έχετε δει δεδομένα δύο μελετών, που ήταν πολύ ακριβές, ε, που δείχνουν ότι ε, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον αυτό, διότι είναι πολύτιμα αλλά και ευάλωτα οικοσυστήματα. Όσον αφορά την ερώτησή σας, εάν υποτιμούμε ε, τον, ε, τα μεγέθη. Θα, ήθελα να σας πω ότι τα δεδομένα αυτά αφορούν οποιονδήποτε έχει εκφορτώσει πάνω από 100 κιλά. Και, στην ομάδα αυτή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μία φορά το χρόνο έχουν αλλιεύσει πάνω από 100 κιλά. Ε, στην ίδια ομάδα μπορεί ε, να υπάρχουν ε, ε, των οποίων το 40% των αλλιευμάτων να είναι αλλιεία βαθαίων υδάτων. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε διαφορετικό κατόφλι 10% των συνολικών αλλιευμάτων σε μια συγκεκριμένη μέρα αλλιείας. Ε, ναι, αν δείτε τα δεδομένα αυτά, ε, λέτε ότι όλους θα επηρεάσουν τα μέτρα αυτά, αλλά ναι, κάποιος μπορεί να επηρεαστεί ε, για το 1 τέταρτο μιας, της δουλειάς μιας ημέρας, ενώ άλλος αλλού μπορεί να επηρεαστεί το 40% των δραστηριοτήτων του. έχουμε... Δεν θέλουμε λοιπόν να καταργήσουμε τελείως τις τράτες ή τα δίχτυα, ε, όλοι θα επηρεαστούν, ε, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Αυτοί λοιπόν που ψαρεύουν με τράτα σήμερα, εάν έχουν σημαντικό μερίδιο τέτοιας αλληλείας, μπορούν να επιλέξουν ε, αλληλευτικά εργαλεία τα οποία να μην επηρεάζονται από την βαθμία κατάργηση. Μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη κατανόηση του τι προτείνουμε. Η κυρία Φράγα ρώτησε εάν η Επιτροπή θα τροποποιήσει την πρόταση. Κυρία Φράγα, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν μπορώ. Ε, αυτή θα είναι απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων. Αλλά μπορώ να σας πω ότι εδώ δίνουμε περισσότερες πληροφορίες και κάνουμε μια εις ανάλυση. Αλλά Η σημασία της πρόταση αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που είναι και παραμένει η ίδια με πριν τρία χρόνια. Εάν όμως ε, υπάρχει ε, θέμα σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε με την πρόταση αυτή, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει το Σώμα των Επιτρόπων. Ε, εγώ δεν έχω εντολή να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα. Κοιτώ τις σημειώσεις μου. Η κυρία Φράγα έκανε κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με τη βελτίωση των ε, αποθεμάτων. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ναι, έχουν βελτιωθεί τα αποθέματα, αλλά είναι γνωστό από τις παρουσιάσεις της ΆΕΣΗΣ ότι αυτά εδώ πέρα επηρεάζουν ε, έναν αριθμό αποθεμάτων πολύ μικρών. Θα επανέλθω στα δεδομένα που σας παρουσίασα ήδη. Σε όλα αυτά τα σκάφη που δηλώνουν τα αλλιεύματά τους. Έχουμε πάνω από, 1.000, από, είδη. Κάποια από αυτά είναι είδη βαθαίων υδάτων, αλλά ο αριθμός των ειδών που καλύπτεται στον κανονισμό είναι 20, 25, 30 είδη βαθαίων υδάτων και από αυτά τα είδη μόνο τα 11 προστατεύονται μετά και ποσοστώσεις. Ε, τα υπόλοιπα δεν προστατεύονται, δεν μελετώνται και δεν αξιολογούνται. Να το έχετε παρακαλώ λοιπόν ε, και αυτό υπόψη κατά τη συζήτησή σας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, ναι, ε, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ε, δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα εντός δύο εβδομάδων. Δεν μιλάμε για μακρύ χρονικό διάστημα, θα έχετε σύντομα τις πληροφορίες που εξετάζουμε. Και αυτά. Νομίζω ότι έκανα όλες τις απαραίτητες διευθύνσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγα για μια διευκρίνηση και μετά ο κύριος Αρσένης. Είπατε ότι τα πλάδια μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα εργαλεία, ασφαλώς. αλλά ας είμαστε σαφείς, ποια είναι η εναλλακτική λύση για το παραγάδι. Ε, οι επιστήμονες μας είπαν ότι το, τα παραγάδια είναι ε, αρκετά πολύ διαδεδομένα ιδιαίτερα σε είδη τα οποία κινδυνεύουν όπως για παράδειγμα οι καρχαρίες μεγάλου βάθους. Ε, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αυτό, διότι αν είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα πολύ μεγαλύτερο, Ε, και μην, μας πει, μην καν ότι το, τα παράδια είναι καλά για τους καρχαρίες γιατί εδώ πέρα ξέρετε την ευαισθησία μας. Μετά, αν αλλάξουμε τα πλάδια με παραγάδια δεν σημαίνει αυτό ότι ορισμένα είδη δεν θα μπορούν να αλλιεύονται. Δηλαδή αλλάζουμε ένα εργαλείο δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε παραγάδια για να ψαρεύουμε τα ίδια είδη. Οπότε για τα είδη δεν πρόκειται να πω τίποτα αλλά αυτό που υπόθηκε είναι ότι τα είδη τα οποία αλλιεύονται κυρίως με τα παραγάδια είναι ε, είδη τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ανάκτησης. Ξέρω ότι υπάρχουν 100.000 είδη, okay. αλλά αυτά κυρίως που θα αλλιεύονται με την αλλαγή του εργαλείου είναι αυτά. Αυτά για να δώσουμε στο κάθε πράγμα την αξία του. Αυτό είπα εγώ. Μην ε, βάζετε στο στόμα πράγματα τα οποία δεν είπα. Ωραία. Ο κύριος Αρσένης. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφή όλα αυτά. Καλώ την Επιτροπή να απαντήσει στις παρατηρήσεις των ε, άλλων Ευρωβουλευτών και να συγχαρώ την ε, Επιτροπή για τη βάση της νέας μελέτης αντικτύπου και να συνεχίσει ε, να εργάζεται. Σημείο 16. Τροποποίηση του κανονισμού 850 του 98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών θα ακούσουμε τον κύριο Νικολέσκου, τον εισηγητή που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι τροπολογίες που προτείνει η Κομισιόν είναι ικανοποιητικές. Πρόκειται για ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων, μέτρα κατεξοδότηση και εκτελεστικά μέτρα. Γνωρίζετε την προβληματική, δεν θα σας τα επαναλάβω. Παρόλα αυτά, κάνω ορισμένες προτάσεις τροπολογίας. Για παράδειγμα, ορισμένα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να υπόκεινται σε ε, κατεξοδότηση πράξης και κάποια άλλα άρθρα, κάποια άλλα μέτρα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι ενώ τα προτείνει η Κομισιόν να είναι. Νομίζω ότι έχετε το κείμενο, περιμένω τα σχόλιά σας. Κυρία Φράγα, το πρόβλημά μου αφορά τροπολογία 4. Μιλάτε για το 1324 για την ισχύ του κινητήρα. Δεν νομίζω όμως ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός αναφέρεται σε αυτό. Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση ε, ε, αλλιές μικρής ε, ε, που αλλιεύει καραβίδες κλπ. Εκεί δεν, έχει, δεν ισχύει το επιχείρημά σας. Οπότε το κείμενο της Κομισιόν θα έπρεπε να παραμείνει ως έχει, εκτός και αν μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ζητάτε τροπολογία. Ο κανονισμός ελέγχου δεν αφορά αυτή την πρόταση. Δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο σημείο του κειμένου του 850. Μετά στην τροπολογία 1 δεν καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικό όσο αυτό που είπα προηγουμένως. Άλλα θέματα, κομισιόν. Ε, Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Φράγα. Πράγματι, ε, υπάρχει ένα άρθρο για την ισχύ, αλλά δεν ξέρω γιατί γίνεται σύνδεση με τον κανονισμό ελέγχου. Θα το σκεφτούμε. Ο συνάλφος μου θέλει να σχολιάσει την νομική πλευρά των τροπολογιών 3 και 5, ή συνάδελφός μου μάλλον. Σε ό,τι φορά το σχέδιο έκθεση έχω ένα σχόλιο για την διάρκεια. Καταρχήν, οι δύο καταξιδότητες πράξεις δεν συμπεριλαμβάνονται, καταρχήν για τις δύο πράξεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ε, στο κατάλογο ε, καταξιδότητες πράξεων της Κομισιόν. Έτσι και αλλιώς ως τώρα ήταν εφαρμοστικές πράξεις και θέλουμε να παραμείνουν έτσι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, διάρκεια για τις κατεξοδότης πράξεις ε, η αρμοδιότητα που δίδεται στην Κομισιόν μπορεί να αρθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιοριστεί στα τρία χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει τρία χρόνια είναι πολύ μικρή περίοδος. Προκειμένου να ε, να τις ε, ε, υιοθετήσουμε και να προφανώς να αναφέρουμε και για την εφαρμογή τους. Ευχαριστώ πολύ κύριο Νικολέσκου. Σε ό,τι αφορά την κυρία Φράγα το σημειώνω. Θα βρούμε μια λύση μαζί. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της Κομισιόν για την διάρκεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων, όλοι ε, θέλουμε αυτή η εκχώρηση να έχει μια λογική διάρκεια. Η Κομισιόν τι, τίνει να ζητά όλο και μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι θέμα υποκειμενικό, θα δω τι θα πούν οι συνάδελφοι. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλο ζήτημα, περνάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης γνώσεις για τη θάλασσα 2020, βελτίωση της χαρτογράφησης του βυθού για αλλιευτικούς σκοπούς. Α, ναι, ναι, προθεσμία, ξέχασα. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 5 Ιουνίου το μεσημέρι. Ε, για το θέμα του κ. Νικολέσκου αυτό. Τώρα, σημείο 17, γνωμοδότηση ε, της κυρίας Νέβες Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα μας παρουσιάσει η κυρία Νέβες Πρόεδρε, καταρχήν μια διευκρίνηση. Δεύτερη φορά εδώ ακούω ότι είναι γνωμοδότηση. Όχι, πρόκειται για ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό και την προηγούμενη φορά υποβλή, ε, παρουσιάστηκε ως γνωμοδότηση, ε, ως ε, για την οποία άλλες επιτροπές, κάποια άλλη επιτροπή θα έχει την ευθύνη επί της ουσίας. Όχι, πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιτροπή που είναι υπεύθυνη επί της ουσίας. Θα το διευκρινίσουμε κυρία Πατράου. Ε, τι να σας πω. Ε, η ΕΜΒΗ εμφανίζεται ως ε, υπεύθυνη επί της ουσίας στα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Θα το διευκρινίσουμε και θα το διορθώσουμε. Για να το λέτε εσείς θα έχετε δίκιο. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Προχωρήστε. Ευχαριστώ πολύ το ανέφερα, διότι φαίνεται, εμφανίζεται για δεύτερη φορά λανθασμένο. Πολύ περισσότερο που δεν θα ανταλλάξουμε ξανά απόψεις ε, για αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε περί τίνος ομιλούμε. Ε, έδωσα, μοίρασα στους συναδέλφους ένα έγγραφο που ακολουθεί την διάρθρωση, τη δομή που σας παρουσίασα την πρώτη φορά που μίλησα για το θέμα αυτό. Ε, καταρχήν ε, μιλώ για το, την πράσινη βίβλο για τη ε, γνώση της ε, για τη θάλασσα 2020 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το, που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2012 το έγγραφο αυτό ε, αποτελεί τμήμα της γαλάζιας οικονομίας ε, που έχει άμεση σχέση με την στρατηγική Ευρώπη 2020 εφαρμοσμένη για τη θάλασσα. Να κάνω μία μικρή παρένθεση για να σας πω ότι η σημασία αυτού του εγγράφου ίσως είναι πιο σημαντική τώρα από ότι στην αρχή όταν είχαμε ξεκινήσει. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά μου, οι τελευταίες συζητήσεις, κατά διάρκεια των τελευταίων συζητήσεων όπου συμμετείχε η κυρία Δαμανάκη, ε, αφιερώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της χαρτογράφησης ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος δόθηκε δηλαδή σε αυτό ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά το μέλλον της αλίας. Συνεπώς θέλουμε να δώσουμε, να προβάλλουμε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα πιο ε, πλατή ακροατήριο και μια πιο πλατιά ε, αποδοχή του εγγράφου. Σας είχα μιλήσει αρχικά για τρία βασικά προβληματικά σημεία επίπεδα. Πρώτον, απόκτηση και διαθεσιμότητα δεδομένων. Δεύτερον, συλλογή και διασύνδεση των δεδομένων. Τρίτον, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων. Καταρχήν θέλαμε να δούμε βέβαια ποια είναι αυτά τα στοιχεία Ε, με την συνεργασία σας, όσοι έχετε απομείνει, ε, θα ήθελα να δούμε αν υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να συλλεχθούν. Εγώ έχω σκεφτεί στοιχεία τα οποία δίδονται από αληφτικά που, είναι, ε, που διαθέτουν VMS ε, στοιχεία προκύπτουν από ηλεκτρονικά ε, ημερολόγια ε, των πλοίων ή ηλεκτρονικά ή μη ηλεκτρονικά, συστήματα, άλλα συστήματα παρακολούθησης των ελεκτικών πόρων, συστήματα μέτρησης αλληλευτικής προσπάθειας, σύνθεση και όγκος ποσότητες των αλλιευμάτων, αλιεύ, συγκεκριμένα είδη αλλιευμάτων, ποσότητε αλλιευμάτων σε συγκεκριμένες ε, ζώνες και περιοχές, ε, τύποι σκαφών, ε, εθνικότητα, λιμένα, το κατα... χωρητικότητα, ισχύ, αριθμό, μέγεθος πληρώματος. Σε ό,τι αφορά ε, την αρτική προσπάθεια αριθμός ταξιδιών, ε, βασικές, βασικά εργαλεία, συγκεκριμένα αλλιεύματα, συγγνώμη, χαρακτηριστικά των, των εργαλείων, αλλά και πιο συγκεκριμένα ε, δεδομένα για τα συγκεκριμένα αλλιεύματα, παρεμπίπτοντα αλλιεύματα, γόνος, όρημα αλλιεύματα, ποσότητες κλπ. κλπ. Ε, με βάση αυτά τα δεδομένα ε, μιλώ για τα τρία ζητήματα τα οποία σας ανέφερα. Πρώτον, δηλαδή, λοιπόν, απόκτηση και διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων. μας ενδιαφέρει να δούμε ποιες είναι οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ενθαρρύνουμε την απόκτηση και διαθεσιμότητα δεδομένων, να εξασφαλίσουμε ε, ισορροπία ανάμεσα στην ε, κυριότητα των στοιχείων και στην χρήση τους. Θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα στα στοιχεία τα οποία, των οποίων η απόκτηση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη από τους φορολογούμενους εν πάση περιπτώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τα οποία θα, και, και στα οποία θα πρέπει η πρόσβαση να είναι πιο πλατιά και να τα διακρίνουμε από τα άλλα δεδομένα τα οποία δεν έχουν χρηματοδότηση ή κρατική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση και στα οποία η πρόσβαση θα είναι πολύ πιο ε, περιορισμένη η πρόσβασή τους θα γίνεται με κατόπιν αδείας του κατόχου των δεδομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα που εφαρμόζεται στην Αλία, εδώ η κατάσταση θα είναι πάλι παρόμοια. Θα κάνουμε και πάλι μια διάκριση ε, τα επίπεδα πρόσβαση, τη δυνατότητα πρόσβαση, ανάλογα με το κατά πόσον ή τα αποτελέσματα τη επιστημονική έρευνα ε, έχουν προέλθει με τη βοήθεια χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από κρατικού ευρωπαϊκού φορεί. Τώρα, τι κίνητρα μπορούμε να παράσχουμε για την απόκτηση περισσότερων δεδομένων. Σε ό,τι αφορά δεδομένα διαχείρισης ε, αλευτικών πόρων, Και εδώ η πρόσβαση θα πρέπει να είναι πλατιά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει είτε την επιστημονική έρευνα είτε τα ίδια τα σκάφη. Ε, σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα, θα άξιζε τον κόπο, πιστεύω, να δεχτούμε ως υποψήφια τη σχέδια, τα σχέδια τα οποία εθελοντικά θα παρέχουν τα δεδομένα τους στους φορείς που ενδιαφέρονται. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο, αυτή η εθελοντική παροχή των δεδομένων ή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας να είναι ένα κριτήριο που θα λαμβάνεται υπόψη θετικά για την επιλογή ε, των σχεδίων αυτών, των επιστημονικών αυτών ε, ε, εργασιών για χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα κίνητρο. Πέραν των κινήτρων μιλούμε και για την εμπιστευτικότητα. Ε, και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. η εμπιστευτικότητα θα πρέπει να είναι ανάλογη με το επίπεδο πρόσβασης, με την ευκολία πρόσβασης. Και θα πρέπει επίσης να συνδυαστεί με τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία, παρουσιάζονται τα στοιχεία. Δηλαδή, σε ε, χαμηλότερους ε, δείκτες ε, απορρίτου ε, ε, τα δεδομένα θα είναι πιο λεπτομερή ε, ενώ όταν το απόρριτο είναι πιο σημαντικό έχουμε ένα υψηλότερο βαθμό χαρακτηρισμού τότε τα δεδομένα θα, να, θα μπορούσαν να είναι λιγότερο λεπτομερή, συγκεντρωτικά, ομαδοποιημένα κλπ. Για παράδειγμα έχουμε απλές παραμέτρους, βασικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να δίδονται με μεγάλη λεπτομέρεια. Όμως οι πιο περίπλοκες παράμετροι, οι πιο ειδικέ παράμετροι που χρειάζεται να ερμηνευθούν και να αναλυθούν επιστημονικά, θα μπορούσαν αυτές οι παράμετροι να δίδονται ως προϊόντα δεδομένων ή δεδομένα επεξεργασμένα ήδη, και, δηλαδή να μην δίνουν τα αρχικά δεδομένα, αλλά το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους. Μετά, ε, συλλογή και διασύνδεση δεδομένων. Εδώ επιμένω σε μια, ε, στην απαραίτητη, στον απαραίτητο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη-μέλη και εντός των κρατών μελών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενοποίησης των, ε, της μορφής των δεδομένων. Θα πρέπει δηλαδή τα δεδομένα να παρουσιάζονται με τρόπο αξιόπιστο ε, και με τρόπο ομοιόμορφο, ε, ενώ θα πρέπει να ελέγχεται και η ποιότητα των δεδομένων και των μεθόδων συλλογής τους να ε, μπορεί να επιβεβαιωθεί. Χρειαζόμαστε επίσης πρωτόκολλα ή κοινά μοντέλα, εναρμονισμένα μοντέλα για τις στρατηγικές δειγματοληψίας και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς επίσης και κοινά ε, format ε, παρουσίασης των δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Επίσης, στο σημείο 2 πάλι, συλλογή και διασύνδεση δεδομένων, θεωρώ ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να αναφέρουν ποια είναι η υπεύθυνη εθνική αρχή για την συλλογή, διασύνδεση και επεξεργασία ε, των ε, δεδομένων, καθώς επίσης και για την παρουσίαση και υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε ο συντονισμός να μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Η επιτυχία μάλιστα αυτού του όλου εγχειρήματο ε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συντονισμό όλων των πηγών δεδομένων σε πρώτο επίπεδο και δεύτερον όλων των φορέων που είναι υπεύθυνε για τη συλλογή, διασύνδεση και ε, παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίτο επίπεδο, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων, θεωρώ ότι για να βελτιστοποιήσουμε ε, τα ωφέλη, θα χρειαστούμε ένα σχέδιο διακυβέρνησης και λειτουργίας που θα εγγυάται την αποτελεσματική συλλογή των δεδομένων μέσω ε, της ε, δημιουργίας στα κράτη-μέλη ενός ε, επιστημονικού περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα είναι και πολύ χρήσιμο για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατήσεων και Δεδομένων να δοθεί ένας ε, ε, μόνιμος ρόλος ε, η... θα μπορούσε η δραστηριότητα Αλίας να αποτελέσει μια θεματική ομάδα ε, του EMODNET δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μια θεματική ομάδα ειδικά για την Αλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θεματική ομάδα για τις ανθρώπινες δραστηριότητε. Ενδεχομένως θα μπορούσε βέβαια σε πρώτο, σε πρώτο επίπεδο η Αλία να ενταχθεί εκεί, αλλά θα προτιμούσα να αφιερωθεί στην Αλία μια ειδική θεματική ομάδα, ένα ειδικό πόρταλ. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το EMODNET θα διαρθρώνεται με την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης της Γης, το GMS. E Τέλος, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δράσης. Χρειαζόμαστε στόχους και προθεσμίες στο πλαίσιο ενός προγράμματος δράσης. Αυτό το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εφαρμοστεί και να αποτελεί εγγύηση συνέχειας και προβλεψιμότητας των δράσεων. Με συγκεκριμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο προπολογισμό. Γιατί συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Κάποια στιγμή έχουμε εκλάμψεις ε, σοφίας με νέα προγράμματα, με νέα σχέδια, αλλά χωρίς να προβλεφθεί η συνεχή τους χρηματοδότηση μέχρι το τέλος. Με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να απαξιώνονται. Συνεπώς χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την συνέχεια, την βιωσιμότητα, μακροπρόθεσμα, διότι αυτό το project έχει νόημα μόνο αν πρόκειται να διατηρηθεί. Δεν θα είχε νόημα να, έχουμε, να έχει μία ημερομηνία γέννησης και μία ημερομηνία θανάτου. Αυτά, ε, εν συντομία <laughs> θα έλεγα, ε, αυτές είναι οι βασικές ιδέες της, ε, ε του κειμένου. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πατράου. Δεν έχει ζητήσει κάποιο βουλευτή το λόγο. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τον υπεύθυνο. Γεια σας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ανάλυση της κυρίας Πατραονέβη. έγινε μια δημόσια διαβούλευση. 240 ενδιαφορόμενοι απάντησαν στο έγγραφο από το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, από την κοινωνία των πολιτών και ερευνητές. Και αυτό που λέτε είναι σε αδρές γραμμές αυτό που έλεγαν και αυτοί θέλουν καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα, στα αλληλευτικά δεδομένα, θέλουν καλύτερη πρόσβαση ε, και ε, σύγκριση των αλληλευτικών δεδομένων με τα υπόλοιπα δεδομένα, για παράδειγμα ε, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια στοιχεία για να είναι πιο αποτελεσματική η αλληλεία ή η δατοκαλλιέργεια. Αναφέρθηκαν σε κίνητρα, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι ή να πιέσουμε ή να έχουμε νομοθεσία ώστε να διαθέτουμε τα στοιχεία ή να δοθούν κάποια οικονομικά κίνητρα προκειμένου να πληρωθεί αυτή η επιπλέον προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να είναι πιο εύκολα διαθέσιμα τα δεδομένα. Οι περισσότεροι προτιμούν τη δεύτερη προσέγγιση, που αν δεν κάνω λάθος είναι αυτή που προτιμάτε κι εσείς, να υπάρχουν κάποια οικονομικής φύσεως κίνητρα, Είπατε όχι απαραίτητο σε σχόλια της κυρία Πατραωνέβες εκτός μικροφώνου. Αλλά νομίζω ότι μεταξύ αυτών που απάντησαν, κυρίως ε, ε, από πλευρά εθνικών κυβερνήσεων, φάνηκε ότι δεν ε, χρειάζονται περαιτέρω υποχρεώσεις, αλλά μάλλον κίνητρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτάσεις για τη δημιουργία κινήτρων Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, το οποίο περιλαμβάνει και προϋπολογισμό για τη συλλογή δεδομένων στην Αλία και για το IMOBNET και πολλά από τα στοιχεία ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατήρησης και Δεδομένων ε, είναι χρήσιμα και για την Αλία αυτοί που απάντησαν στη διαβούλευση ήθελαν να συγκεντρωθούν κάπου όλα αυτά τα στοιχεία. Αναφερθήκατε ε, και εσείς στο ενδεχόμενο μιας δικτυακής πύλης για την αλληλεία συγκεκριμένη. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και στη διαβούλευση. Προφανώς λοιπόν και θα το εξετάσουμε και αυτό. Τώρα, τι θα θέλαμε να κάνουμε τώρα μια αξιολόγηση αντικτύπου για να δούμε λίγο τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις και το πρόγραμμα δράσης ε, θα ακολουθήσει. Το πρόγραμμα δράσης είναι ο δικός χάρτης όπως θα τον αποκαλούσε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου το ένα είτε το άλλο, δεν έχει σημασία, τον ίδιο στόχο επιτελούν. Οι εναλλακτικέ λύσεις είναι να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρατε κι εσείς, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα αλευτικά δεδομένα, πώς μπορούμε να τα εξετάσουμε από κοινού με άλλα δεδομένα, και υπήρχε και μεγάλη διάθεση από πλευρά ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν και αυτοί περισσότερο. Όχι μόνο του αλλιευτικού τομέα, αλλά και τη αιωλική ενέργειας ή άλλων αντίστοιχων τομέων και αυτοί θα ήθελαν να συμμετέχουν. Και αναφερθήκατε και στη διακυβέρνηση. there was a lot of Συζητήθηκε πολύ το θέμα της διακυβέρνησης και αναφέρθηκε και κάποιος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα στη διακυβέρνηση. Και αυτό θα αποτελούσε κίνητρο ώστε να νιώσουν ότι συμμετέχουν στην όλη πρωτοβουλία και να μην προστατεύουν τόσο τα δεδομένα. Βεβαίως ε, πρέπει να υπάρξει ε, προστασία στο θέμα της εμπιστευτικότητας. Ε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να είναι απόρριτα τα στοιχεία. Παραδείγματο χάρη θέματα προστασίας για κάποια είδη τα οποία είναι σε κίνδυνο και δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ακριβώς που βρίσκονται για λόγους ασφαλείας και ούτω ε, σε γενικές γραμμές όμως ε, υπάρχει μια κίνηση προς ε, πιο εύκολα διαθέσιμα δεδομένα, πιο ανοιχτά σε όλους. Τώρα, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι εθνικοί φορείς το μοντέλο δεν είναι μια μεγάλη βάση δεδομένων. Ε, κάθε κράτος έχει τα δικά της δεδομένα και διατίθενται ώστε να μπορεί κάποιος να τα δει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή κάποιος που εξετάζει τη βάση δεδομένων μπορεί να δει όλα τα στοιχεία, ε, στοιχεία για τα αλλιεύματα, για παράδειγμα τα αλλιευτικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας, μπορεί να πάρουν στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο και το καθεξής, χωρίς να μην χρειάζεται να δει την κάθε χώρα ξεχωριστά. Ε, τώρα, προτυποποίηση, αναφερθήκατε και σε αυτήν φυσικά. Είχε γίνει κάποια πρόοδο ε, στον τομέα αυτό με τα λευτικά δεδομένα και άλλα δεδομένα. Σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να είναι και ε, δυνατή η χρήση των ελευτικών δεδομένων με άλλα δεδομένα. Σαφώς δεν θέλουμε να είναι μια απλή σπίθα, πρέπει να είναι μια συνεχής ε, διαδικασία. Αλλά στις πολιτικές δημοσιοποιητικές προοπτικέ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας για το 2014-2020 περιλαμβάνεται πρόταση για προϋπολογισμό ε, άρα είναι στα, ε, στις προοπτικές μας. Α, Αναφερθήκατε και στα διαφορετικά επίπεδα δεδομένων. Το σκεπτικό μας είναι ότι ο φορολογούμενος, το κοινό, πληρώνει πολλά δεδομένα και θα πρέπει τουλάχιστον τα βασικά δεδομένα να είναι δημόσιο αγαθό. Εάν κάποιος θέλει πιο εξειδικευμένα δεδομένα για ειδικό σκοπό, τότε θα πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος Και μέσω διάθεσης των δεδομένων δημιουργούνται και κίνητρα για καινοτομία. θα μπορούσαν για παράδειγμα διάφοροι φορές ε, να χρησιμοποιούν τα ελευτικά δεδομένα για άλλες υπηρεσίες, για νέους σκοπούς, για να βοηθήσουν τις αλληλευτικές αρχές αλλά και τους ίδιους τους αλληλείς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα με πρότυπο τρόπο, αλλά Εξαρτάται βέβαια και από το τι ακριβώς εννοείται με ε, διάφορα επίπεδα δεδομένων. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο ε, επίπεδο δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα σε όλους. Για παράδειγμα τα είδη των ειζημάτων στον βυθό της θάλασσας. Αλλά ε, ίσως θα έπρεπε να γίνεται και μία αξιολόγηση στα δεδομένα για να δούμε εάν ε, μπορούμε να προσφέρουμε και αυτό ως υπηρεσία επιπλέον. Ολοκληρώνοντας, Νομίζω ότι αυτά που μας λέτε ε, είναι προς την ίδια κατεύθυνση του δικού μας του σκεπτικού, είναι προς την ίδια κατεύθυνση ε, αυτών που ε, λένε και τα στοιχεία της διαβούλευσης. Ε, καλό θα ήταν να γίνει μια εκτίμηση επιπτώσεων και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα δράσης. Και σημειώνω και το χρονοδιάγραμμα, ακόμα το συζητούμε. Oh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέπαν. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο κύριε Πατρά. Uh, uh, Δύο ερωτήσεις νομίζω. Μιλήσατε για τις μελέτες αξιολόγησης ε, αντικτύπου. Αλλά δεν ξέρετε πότε θα γίνουν ακριβώς. Μήπως θα μπορούσα να τη δω αυτή την έκθεση πριν ε, ολοκληρώσω την έκθεση. Δεύτερον, ίσως δεν σας κατάλαβα καλά, αλλά μιλήσατε για πληρωμή για την πρόσβαση των δεδομένων, ότι τα πιο βασικά, τα πιο θεμελιώδη δεδομένα θα είναι δωρεάν, διαθέσιμα, αλλά πιο ειδικά δεδομένα θα πρέπει να, ε, ε, να είναι επιπληρωμή η πρόσβασή τους. Σας κατάλαβα καλά. First question, the impact... Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η μελέτη επιτύπου θα διατεθεί. Θα πρέπει να κοιτάξω τις ημερομηνίες με την υπηρεσία μου. Ε, σας παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεται ε, ο συνάδελφός σας που πληκτρολογεί στον, υπολογιστή δίπλα. Before we do... Ωραία. Πριν εκπονήσουμε τη μελέτη αντικτύπου θα δημοσιευθεί ο δικός χάρτης για τη μελέτη αντικτύπου. Και μετά θα έχουμε άλλον έναν οδικό χάρτη, το ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε τη μελέτη αντικτύπου όταν ολοκληρωθεί. μάλλον θα ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι, πιστεύω. οτιδήποτε χρηματοδοτηθεί από το EMFF ε, θα ε, δημοσιευτεί, θα είναι προσβάσιμο χωρίς χρέωση. Εάν άλλοι θέλουν ε, να παρέχουν προστιθέμενες πρόσθετες υπηρεσίες με βάση τα δεδομένα αυτά, είναι δικό τους θέμα αν θα τις χρεώσουν ή όχι. Εάν κάποιο θέλει να οργανώσει δηλαδή κάποια ειδική υπηρεσία για του αλληλεί ή τι ε, αλληλευτικέ αρχέ, ε, κάτι που θα του ε, στοιχήσει χρόνο, μπορούν να το χρεώσουν. Αλλά ό,τι προέρχεται από εμά θα είναι δωρεάν. Πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Δεν έχουμε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί στι 9. Πρόεδρε, ευχαριστή τη Ερμηνεία. Ευχαριστούμε και εμεί. Εσά αύριο το σπουδαίο.